Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, προσκεκλημένοι μας. Κυρίες και κύριοι, ξεκινούμε τη δημόσια ακρόαση για την νομοποίηση παρανόμων εσόδων, ε, παρεμβάσεις της Ρωσίας και συνέπειες αυτής ε, στα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την εταιρεία Tax 3. Έχουμε λοιπόν τα εξής πάνελ. Στο πρώτο συζητούμε τις συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση των περιπτώσεων νομοποίησης παράνομων εσόδων που έχουν συνάφεια με παράγοντες από τη Ρωσία. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ομιλητές από το πρώτο πάνελ, τον κύριο Άντερς Οσλούντ. Καλώς ήρθατε. Στο Ατλαντικό Συμβούλιο και στο Georgetown University καθηγητής θα μας μιλήσει για την νομοποίηση παρανόμων εσόδων... από τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς έχει καταστεί αυτό ε, απειλή για την εθνική ασφάλεια στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γιώσουα Κίρκενμπαουμ είναι ο επόμενος ομιλητής. Καλώς ήρθατε από, το, από τη συμμαχία του γερμανικού σχεδίου Μάρσαλ και ασχολείται με την ε, παράνομη χρηματοδότηση. Έχει συντάξει μάλιστα ένα έγγραφο που, όπου προτείνει μια καλύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για την νομοποίηση των παρανόμων εσόδων. από την αντιπροσωπεία τη ΤΑΞΤΡΙΑ 3 είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον κύριο Κίρχενμπαουμ στην Ουάσιγκτον ε, ε, τον προηγούμενο μήνα, μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Θα ήθελα επίση να καλωσορίσω τον κύριο Ρίτσαρτ Μπρούξ, δημοσιογράφο του Private Eye και του Guardian. Έχει μελετήσει και διερευνήσει αρκετές υποθέσεις νομοποίησης παρανομών εσόδων από τη Ρωσία. Θα έχετε μέχρι 7 λεπτά ο καθένας για τις εισαγωγικές σας ομιλίες και παρακαλώ τον κύριο Όσλουντ να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, αυτή την για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα η νομοποίηση παρανόμου χρήματος από την Ρωσία αποτελεί κατά την άποψή μου σημαντική απειλή για την εθνική ασφαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και πρέπει να αναλυφθούν αμέσω μέτρα κατά αυτής της μάστιγας. Η πρώτη θεραπεία λοιπόν θα ήταν η οικονομική διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχώς έχει αναλάβει τα κατάλληλα βήματα για την αντιμετώπιση με την ε, οδηγία το 2018 τον Ιούνιο για την καταπολέμηση των παρανόμων εσόδων. Οι κύριες διατάξεις αυτής της οδηγίας προβλέπουν ότι σε όλα τα από όλα τα κράτη-μέλη απαιτείται να εξασφαλιστεί πως οι πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο κάθε νομικού προσώπου θα είναι προσβάσιμες στις αρμόδιες αρχές και σε οδήποτε μέρος του ευρέως κοινού ή των πολιτών. Είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί πλήρως αυτή η οδηγία. Θα ξεκινήσω αμέσως με τη φύση του τωρινού καθεστώτος της Ρωσίας υπό τον πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν. Έχει προχωρήσει προς ένα αυταρχικό καθεστώς και κράτος η Ρωσία ε, όχι μόνο όμως αυταρχικό αλλά και αυταρχική κλεπτοκρατία. Το καθεστώς του Πούτιν ε, ε, ισούται με την συγχώνευση της ασφάλειας των αστυνομικών αρχών ασφάλεια και του οργανωσμένου εγκλήματος. Δηλαδή δεν πρόκειται για ένα κράτος το οποίο λειτουργεί κατά τρόπο κανονικό, αλλά ένα κράτος το οποίο λειτουργεί προκειμένου να εμπλουτίσει και να δώσει περισσότερη εξουσία στην ηγεσία. Έχω μάλιστα μία μελέτη με το βιβλίο «Ο καπιταλισμός ε, το, της ηγεσίας της Ρωσίας και το η πορεία, το μονοπάτι από την οικονομία της αγοράς στην κλεπτοκρατία που έχει εκδοθεί από το University Press της, ε, του Yale το Μάιο του 2019 όπου αναφέρομαι στο κράτος, τις κρατικές εταιρείες και τους ακολούθους του Πούτιν ε, που αντλούν πόρους από το κράτος και τις επιχειρήσεις τους. Επιχειρήσεις του. Με απόλυτη αποφασίωση στον Πούτιν όλοι αυτοί. Ε, από την, μεγάλη, από την Αγία Πετρούπολη. Ε, έχουν εργαστεί με τον Πούτιν για χρόνια. Δεν προέρχονται όλοι από το ΚΑΚΕΜΠΕ γιατί η αφοσίωση στον Πούτιν είναι πολύ πιο σημαντική από την προέλευση από την ΚΑΚΕΜΠΕ Και έτσι έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικό καθεστώς, ένα καθεστώς το οποίο έχει φτάσει πλέον να μην ελέγχεται καν από τον ε, Πούτιν. Έτσι λοιπόν είναι τεράστιες οι συνέπειες αυτής της κλεποκρατίας. Από το 2004 ο Πούτιν και οι πιο στενοί φίλοι του έχουν αποσύρει μόνο από την Κάσπρο 10 έως 15 δισεκατομμύρια ε, δολάρια για προσωπικό κέρδος. Όχι για να το επενδύσουν στο κράτος, αλλά για να μοιραστούν το, το ποσό αυτό 4-5 άνθρωποι και 15 έως 25 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν αυτά τα οποία έχουν αντιληφθεί από το ρωσικό κράτος και τις κρατικές επιχειρήσεις συνολικά από το 2006. Η τραγική ηρωνία είναι ότι τα χρήματα αυτά δεν μπορούν καν να τα κρατήσουν στη Ρωσία γιατί η Ρωσία δεν γνωρίζει κράτος δικαίου και ως εκ τούτου δεν αισθάνονται ότι είναι ασφαλή τα δικαιώματα ιδιοκτησίας πάνω στα ποσά αυτά και άρα αναγκάζονται να τα εξαγάγουν. Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε με στοιχεία τεκμηριωμένα που μας δίνουν τα πρόσωπα Γκενάντι Τιμσένκο, Αρκάντι Ρότεμπερκ, τον αδελφό του Μπόρις Ρότεμπερκ και τον Γιούρι Κόβαλτσουκ που είναι όλοι παλιοί φίλοι του Πούτιν από την ε, Αγία Πετρούπολη. Και οι τέσσερις αυτοί έχουν ε, καταδικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις μόνο κατά του Αρκάντι Ρότεμπεργκ και του Γιούρι Κόβαλτσου, γιατί ο Τιμτσέγκο και ο Ρότεμπεργκ και ο Μπόρις Ρότεμπεργκ είναι Φινλανδοί υπήκοοι και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Ένωση, Φινλανδοί είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Επίση, έχει πολύ στενή συνεργασία, έχουν πολύ συνεργασία με το Κρεμλίνο, προσφέροντα ε, πολλαπλέ υπηρεσίε ε, αυτοί οι άνθρωποι. Ιδιαίτερα ο Αμπράμοβιτ, αλλά και ο Ντεριπάσκα, ο Ουσμάνοφ, ο Κερίμοφ είναι τα πιο προφανή παραδείγματα ολιγαρχών του Κρεμλίνου κατά των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ μόνο και μόνο κατά τον Τεριπάσκα και Κερίμοφ και κατά κανένας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι υπεύθυνη για την ε, απώλεια έως και 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την περίοδο του 1999 από τη Ρωσία, χρήματα τα οποία έχουν κρύψει Ρώσοι υπήκοοι στο εξωτερικό. Τεράστιο ποσό. Η πορεία των χρημάτων αυτών περνάει μέσα από την Κύπρο λόγω του η συμφωνίας ε, περί μη διπλής φορολογίας μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ρωσίας του 1982. Και στη συνέχεια τα χρήματα προχωρούν προς τα νήσου Βέρτζιν του Ηνωμένου Βασιλείου, τα, τις Κέιμαν και από εκεί στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα στο Wilmington και το Delaware. Και από εκεί συνεχίζουν. με επενδύσεις στη συνέχεια σε ακίνητα στο μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης έχουμε ιδιωτικά ταμεία επενδύσεων, hedge fund και συστήματα μετοχικά στις ΗΠΑ, Πολιτείες που περνούν, όπου περνούν τα ποσά τελικά στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Και μια και περνάει ο χρόνος, θα προχωρήσω απευθείας στις, ε, συμπεράσματά μου. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιβάλλουν προσωπικές κυρώσεις κατά των ακολούθων του Πούτιν και των ολιγαρχών που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Κρεπλίνου στο, από το εξωτερικό, φίλους του Πούτιν ε, συγγενείς ε, εκείνων που διακρατούν κεφάλαια για λογαριασμό του Πούτιν. Ο Πούτιν έχει αποδείξει ότι ανταποκρίνεται μόνο σε προσωπικής φύσης κυρώσεις. Και γι' αυτό και ο νόμος Μαγνίτσκι έχει τόσο μεγάλη σημασία. Όπως άλλωστε και οι προσωπικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στους πιο στενούς του φίλους. Και έτσι προχωρώ στη σύσταση ότι θα πρέπει τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν νομοθεσία αντίστοιχη με, την, νόμο Μαγνίτσκι, με το Μαγνίτσκι Act και να την εφαρμόσουν. Στόχος είναι η διαφάνεια. Αφενός μεν ως προς την αναγνώριση του πραγματικού και τελικού ιδιοκτήτη αυτών των κονδυλίων που θα πρέπει και να δημοσιοποιείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την οδηγία για την καταπολέμηση των παράνομων εσόδων και δεύτερον θα πρέπει όλοι οι δημόσιοι ε, το, προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών και δημόσιοι υπάλληλοι να κάνουν δηλώσεις ποθενέσχες, δημόσιες όπως άλλωστε γίνεται και στις χώρες του Βορρά της Ευρώπης από το 18ο αιώνα. Γιατί πολλοί πρώην πολιτικοί, οι αξιωματούχοι, οι πρώτης γραμμής επιχειρηματίες έχουν με νόμιμο τρόπο αποκτήσει θέσεις σε διοικητικά συμβούλια ή συμβουλευτικές θέσεις σε μεγάλες ρωσικές εταιρείες. Ο Γκέρχαρτ Σρόντερ είναι το πιο χτυπητό παράδειγμα του πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Και βέβαια όλοι αυτοί δείχνουν απόλυτη αφοσίωση και πρέπει να το καταγγείλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καθηγητή. Σας ευχαριστούμε για την εισαγωγή σας, η οποία έδειξε ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα θέμα παγκόσμια εμβέλεια. Ο κύριο Κίσενμπαουμ έχει τον λόγο τώρα. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή, σα ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημαντική ακρόαση. Ε, με μεγάλη τιμή και χαρά εμφανίζομαι στην Επιτροπή σα. Οι παράνομε οικονομικέ δραστηριότητε από τη Ρωσία και την κοινωνία ανεξαρτών κρατών είναι ένα θέμα που πρέπει να μπει ψηλά στη διμερή ατζέντα Ευρωπαϊκή Ένωση Αμερική. Τα πρόσφατα χρόνια ε, υπάρχουν πολλοί άριθμα σκάνδαλα ξεπλήματος χρήματος στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Ε, δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλένονται μέσω ενό ε, φορέα. Ε, οι συχνοί δεσμοί με την ΚΑΚ και με τη Ρωσία ανεπαρκεί πρόστιμα απουσία ποινικών διώξεων. Ακόμα και όταν αυτά τα συστήματα έχουν σαν σκοπό τη διευκόλυνση τη διαφθορά ή τη εγκληματικότητα εκεί πέρα, δηλαδή στη Ρωσία, η ανοχή αυτών των δραστηριοτήτων εντό Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί κινδύνου εδώ πέρα. Τα επαγγελματικά δίκτυα διευκόλυνση, τα οποία ελέγχουν αδιαφανή κανάλια και τις χρησιμοποιούν για καλούς εντός αγωγικών σκοπούς ε, ροής, ροές κεφαλαίων, α πούμε, συχνά προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτούς που θέλουν να κάνουν πολιτικές παρεμβολές στα κράτη-μέλη. Το να επιτρέπουμε στις ε, τράπεζες και σε άλλους να έχουν ε, δραστηριότητες που βασίζονται σε αδιαφανή ή παράνομα κονδύλια από την ΚΑΚ, δημιουργεί προβλήματα γιατί δημιουργεί χώρους ανοιχτούς και ευάλωτους στη ρωσική πολιτική οικονομική επιρροή. Επιπλέον, ε, η ρωσική επιρροή μπορεί να, αντικαταστεί, να αντικατασταθεί από απρόβλεπτες γεωπολιτικές δυναμικές στο μέλλον. Αυτά τα σκάνδαλα, συχνά αλλά όχι πάντα, επικεντρώνονται στα μικρότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, που έχουν όμως μεγάλους ε, τραπεζικούς τομείς offshore. Η εποπτεία για το για την καταπολέμηση του ξεπλήματος του χρήματος είναι επαρκής σε χώρες όπως η Κύπρος, η Λετωνία, όπου έχουμε πολλές δραστηριότητε, αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εφαρμόζεται επαρκώ ε, το δίκαιο περί ε, καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος του χρήματος. Ένα σύστημα όπου οι τράπεζες δέχονται πρόστιμα λίγων εκατομμυρίων ευρώ για παράδειγμα δραστηριότητε δισεκατομμυρίων ευρώ θα αποτύχει η, επιδεινώνεται το πρόβλημα της ε, επαρκούς ε, εφαρμογής ε, λόγω του ότι η εποπτεία για το ξέπνο του χρήματος είναι εθνική δραστηριότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η αδειοδότηση και όλες οι εγκρίσεις που δίνονται είναι της εμβέλειας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χωρίς σωστό μηχανισμό εποπτείας ε, στην Ευρωζώνη και ενώ οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αυτές παίρνουν ε, το διαβατήριο για να παρέχονται σε ολόκληρη την ε, ενιαία αγορά. Ε, συμφωνώ λοιπόν με την Ντανιέλ Νουγή του, Ευρωπαίου, του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας και τον Μπενουά Κιωρέ του Συμβουλίου της ΕΚΤ και υποστηρίζω μια κεντρική αρχή που να ασχολείται με την με τον έλεγχο του ξεπλήματος του χρήματος. Η υπηρεσία αυτή θα εποπτεύει τις τράπεζες και τους μη τραπεζικούς φορείς ε, σε όλη την ενιαία αγορά, θα είναι ανεξάρτητη πολιτικά, θα έχει μοναδική πραγματογνωμοσύνη και θα εφαρμόζει, ε, θα έχει εξουσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ισχυρή κεντρική υπηρεσία θα είναι δραστήρια, θα είναι πολιτικά ανεξάρτητη και θα έχει πραγματικά ε, τον πρώτο λόγο στον χώρο αυτό. Θα χρησιμοποιεί δεδομένα, ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες ε, εποπτικές αρχές και θα μπορεί να εκδίδει ε, πολύ αποτραπτικά και έντονα δάνεια, ε, ε, συγγνώμη, πρόστιμα, ε, για όσους παρανομούν. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε και άλλες ε, αρχές για να... Όλα αυτά μάλλον μπορούν να γίνουν υπό το σημερινό ε, πλαίσιο. Φυσικά οι τράπεζες ε, παίζουν ένα μοναδικό ρόλο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα εστιάσω στο ρόλο των τραπεζών. Είναι ένα μια μεγάλη πρόκληση, αλλά όχι το μόνο πρόβλημα. Έχουμε τώρα την οικονομική τεχνολογία ε, συχνά όλε οι δραστηριότητε αυτέ γίνονται εκτό του επίσημου τραπεζικού συστήματο, ε, και αυτό δείχνει τη σημασία τη ισχυρή εποπτείας όταν μεταφέρονται οικονομικά ποσά, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, η διαπραγμάτευση κινητών αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική, είναι μια δραστηριότητα λιγότερο διαφανής ε, από την είναι οι διεθνεί ε, πληρωμές που γίνονται από τις τράπεζες. Ε, και συχνά δεν ξέρουμε του πραγματικού δικαιούχου. Ο Λουί Δεκίντο, αντιπρόεδρο τη ΕΚΤ, ε, προειδοποίησε ότι οι δραστηριότητε αυτέ έχουν μεταφερθεί από τι ε, τράπεζε σε επενδυτικά ταμεία, σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, σε αμοιβά κεφάλαια τη άθμιση κινδύνου και εδώ έχουμε του συστημικού κινδύνου. Οι παράνομοι φορεί μπορούν να προσπαθήσουν να χωθούν σε αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια ε, και να, ε, γιατί ελκύονται από την έλλειψη διαφάνειας ε, και την πολύ ελαφριά και ανεπαρκή εποπτική δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει ποιε είναι οι προτεραιότητέ τη. Να εποπτεύει τι τράπεζες, θα πρέπει να αξιολογήσει και την εποπτεία αυτών των ιδιωτικών επενδυτικών ταμείων κτλ. Η, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προσπάθειες ε, να τηρήσει τα διεθνή πρότυπα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εδώ και 17 χρόνια ε, καθυστερεί να εφαρμόσει τα διεθνή πρότυπα σε αυτόν τον τομέα. Το, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η έλλειψη διαφάνειας στις επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι ΗΠΑ, δεν ξέρουν ποιος επενδύει, ε, σε τι, που βρίσκεται και γιατί κάνει αυτές τις επενδύσεις οι κυβερνήσει ε, έχουν ε, μία ανοιχτή στάση για τι επενδύσει, αλλά απλώ δεν ξέρουν ποιο ε, κατέχει τι. Πιστεύω ότι αυτό το περιβάλλον οδηγεί κρατικού ή μη κρατικού φορεί από αυταρχικέ χώρε όπω η Ρωσία αλλά και άλλε να δημιουργήσουν μεγάλε και ισχυρέ στρατηγικέ επενδυτικέ θέσει χωρί να δίνουν στοιχεία στι ελεγκτικέ αρχέ, στι εποπτικέ αρχέ ή στι διοκτικέ αρχέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει πρόσφατα πιο σωστές ε, διαδικασίες εποπτείας. Ε, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια ε, για τις άμεσες επενδύσεις και για το, τις εταιρείες χαρτοφυλακίων, ούτως ώστε οι ελεγκτικές αρχές και οι διοκτικές αρχές να ξέρουν πολύ καλά που πηγαίνουν οι πόροι ε, μεγάλης αξίας. σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ΗΠΑ. Ε, πιο επιθετική στάση με ποινικέ διώξει ε, ε, των παράνομων αυτών ε, ενδιάμεσων των τραπεζιτών και των παρόχων επαγγελματικών υπηρεσιών θα έχουν τεράστιο αποτρεπτικό χαρακτήρα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε καταδικαστικές αποφάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να συνεχίσουμε όμως τις προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. κύριος Μπρούξ τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα σε μια σημαντική συγκυρία. Βλέπουμε ότι το θέμα της διεθνούς διαφθοράς αποτελεί πλέον πολιτική απειλή. Διεθαρμένα πολιτικά συστήματα όπως το ρώσικο συντηρούνται από την κλοπή και το ξέπλυμα χρήματος και έτσι μπορούν να υπονομεύουν την δημοκρατία αλλού όπως είδαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Οπότε ε, αυτό το οποίο ήταν ε, εγχώριος κίνδυνος ε, για τις χώρες που διαγούμιζαν η ελίτ τώρα μας επηρεάζει όλους. Και βεβαίως έχουμε και τα αποτελέσματα της κρίσης που μας καθιστούν πιο ευάλωτους σε αυτές τις απειλές όπως δείχνει το Brexit και βεβαίως αυτό φέρνει μαζί του και την λιτότητα που έχει και αυτή τα δικά της προβλήματα δηλαδή το κλειδί είναι οι πληροφορίε. Πρέπει να γνωρίζουν οι διοικητικές αρχέ που πηγαίνουν τα λεφτά, αλλά οι πιθανότητε να συμβεί κάτι τέτοιο είναι πολύ χλωμέ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματο χάρη το 2007, όταν ήταν λιγότερο σοβαρή η απειλή, η τότε κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει το προσωπικό τη αρμόδιας υπηρεσία από 100 στου. 200 τελικά έμειναν 80 και έχουν 400.000 περιπτώσεις να ερευνήσουν κάθε χρόνο. Μόνο μετά την επίθεση στο Σόλσμπερι έχουν αφιερωθεί επιπλέον πόροι. Δεν θα μπω τώρα στους αριθμούς, αλλά εκτιμάται ότι το ξέβλημα χρήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γύρω στα 90 δισεκατομμύρια λίρες, γύρω στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάει η κυβέρνηση. Και για αυτά βεβαίως ε, ξοδεύουμε γύρω στα 100 εκατομμύρια λίρες ε, στον τομέα της εποπτείας. Βεβαίως έχουμε ένα πολύ μεγάλο τραπεζικό τομέα αλλά και πάρα πολλές χιλιάδες εταιρείες γράμματοκιβώτια και ΕΠΕ που μπορούν να υποβάλουν ψεύτικα νούμερα με ατιμορρησία. Αυτά τα σχήματα είναι το κύριο μέσο ξεπλήματος ε, χρήματος όπως έχει αποκαλύψει απατηχέρμητα και άλλες. Αλλά Έχουμε γύρω στα 4 εκατομμύρια εταιρείε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το δε μητρό έχει 20 άτομα προσωπικό για να τις ελέγχει. Οπότε έχουμε δει κάποιες χρήσιμες νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες, ε, νομοθεσίες ε, για τον Μαγνίτσκι, αλλά και νομοθεσία η οποία επιτρέπει την δίμευση με αστική διαδικασία αγαθών που δεν ε, δικαιολογούνται. Αλλά αυτό είναι περισσότερο πολιτικό ζήτημα. Μέχρι στιγμής μόνο μία τέτοια εντολή έχει εκτελεστεί σε ένα έτος που βεβαίως ε, χαροποίησε ιδιαίτερω τι εφημερίδες γιατί αφορούσε διαμάντια και αγορές 60 εκατομμυρίων λιρών στα Χάροτς αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά αυτά τα εργαλεία. Και βεβαίως η ποινική πλευρά οι ποινικέ κυρώσεις είναι ακόμη πιο καταθλιπτικές ως εικόνα. Δεν γνωρίζω να υπάρχουν κάποια χρήματα από τις πρώην Σοβιετικές χώρες ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο που να κατέληξαν σε ποινική δίωξη. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μία πρόσκληση για να ξεπλύνουν τα χρήματά τους. Στην απίθανη περίπτωση που θα γίνει κάτι, ουσιαστικά θα είναι ένα μικρό κόστο σε σχέση με τον όγκο των χρημάτων. Εδώ και χρόνια εγώ και άλλοι παρακολουθούμε τα χρήματα που μπαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κυρίως αρκετά από αυτά πηγαίνουν και σε ακίνητα του Λονδίνου και μιλάμε για μια αγορά 4 δισεκατομμύριων λιρών το έτος, ένα έτος και μετά υπάρχουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες, τα ιδιωτικά σχολεία και τα σχετικά. Και παρουσιάζουμε κάπου αυτήν τη δραστηριότητα. Και ε, έχουμε και την οικογένεια του πρώην δημάρχου της Μόσχας που έχει μια, ένα μέγαρο στο Κένζιγκτον και ενώ οι μεγάλες αγγλικές τράπεζες ε, μάλλον έχουν απομακρυνθεί από αυτό το φαινόμενο, οι μικρότερες ε, εξακολουθούν. Υπάρχει μια τράπεζα στο Mayfair ονόματι EFG που αγόρασε την Κούτς και μεταξύ άλλων ε, δέχτηκε 100 εκατομμύρια δολάρια από έναν φίλο του Τσετσένου πρόεδρου. Και βεβαίως ο πρόεδρος της τράπεζας ε, είπε ότι αν και δεν του αρέσει ιδιαίτερο, είναι προαπαιτούμενο για να έρθουν και άλλοι πελάτες. Δεν φαίνεται να τον ανησυχούν ιδιαίτερα τα φαινόμενα ξεπλήματος χρήματος. Βεβαίω, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά γρήγορα με το να έχουμε περισσότερους ε, πόρους, γιατί και οι διοκτικέ αρχές δεν έχουν τις ε, ικανότητε και την εμπειρία και οπωσδήποτε στον Βασίλειο και υποψιάζομαι και αλλού υπάρχει τεράστια δουλειά που πρέπει να γίνει και θα αργήσει. Έχω την εντύπωση πως θα πρέπει να δούμε την ε, διεθνή διαφθορά όπως βλέπουμε την φτώχεια και τις ε, αρρώστιες. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή εξοδεύει 0,7% του ΑΕΠ του για την ε, διεθνή ανάπτυξη ενώ για την καταστολή του εγκλήματος έχει ένα 0,04% του ΑΕΠ. Βεβαίω, μιλάμε για ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο περιλαμβάνει εταιρείε λογιστών και δικηγορικά γραφεία. Η έκθεση που σας ε, απέστειλα δείχνει διάφορους ε, τομείς ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα οι τράπεζες έχουν βοηθηθεί από τους λογιστές τους και κατ' επανάληψη κάνουν τα στραβά μάτια ακόμα και σε περιπτώσεις όπου έχουμε τόσο ενδυμικό ξέπλυμα χρήματο που θα πρέπει να το έχουν παρατηρήσει και θα πρέπει βεβαίως είναι στα καθηκοντά τους να το επισημάνουν και στις αναφορές που δίνουν στις ρυθμιστικές αρχές. Μιλάμε για μεγάλες ε, εταιρείε λογιστικές, τις μεγάλες ε, που συνεχώς μας μιλάνε για εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ιδιαίτερο στι βαλτικέ χώρες. Η Ernst Young ε, που έχει σύνθημα ότι φτιάχνουμε έναν καλύτερο κόσμο συχνά έχει δεχθεί καταγγελίε ε, στα κεντρικά της, στο Λονδίνο Λοιπόν, έχει δεχθεί επώνυμες ε, καταγγελίες. Είδε PMG όταν ήταν η Λετωνία στην ε, μόδα είχε επίσης μεγάλο ρόλο εκεί. Η Deloitte ε, πώς δεν πρόσεξε τα 200 δισεκατομμύρια ξεπλήματος στην Danske Bank. Βεβαίω, οι ίδιες εταιρείες συνεχίζουν να σφραγίζουν τους λογαριασμούς των εταιριών στην Μόσχα και βεβαίως αυτό είναι το πρώτο βήμα της διαφθοράς αν δεν τους διατάξει το Κρεμλίνο, όπως έγινε με την Γιούκος πριν από 10 χρόνια, πότε δεν φέρνουν καμία αντίρρηση για τα νούμερα. Ο κ. Άσλοντ μόλις ανέφερε τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την Gazprom, δηλαδή τους ξέφυγε στην PwC. Λέω στην έκθεσή μου το πόσο κοντά είναι στο καθεστώς οι παγκόσμιες αυτές εταιρείε ε, μέσω των συνεδρίων κτλ η ηγεσία τους ε, δεν βγαίνει στη σύνταξη και πάει στα ΔΣ των εταιριών αυτών που συνδέονται με το Κρεμλίνο. Και οι δικηγόροι επίσης ε, μεγάλο δικηγόροι που ε, εμπλέκονται σε αυτές τις αγορές ακινήτων εκατομμυρίων λιρών. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε δει παραδείγματο χάρη τα πόθεν έσχες Ρώσων βουλευτών όπου βλέπαμε κάποιον άνθρωπο να αγοράζει ε, διαμερίσματα στο Λονδίνο χωρίς να έχει κανένα εισόδημα. Τέτοια λοιπόν ε, δικηγορικά γραφεία δρούν για λογαριασμό ολιγαρχών που έχουν μάλλον ύποπτο πλούτο. Και ε, βεβαίως η κρίση τους επηρεάζεται και από το τι είναι υποφελές για τους ίδιους. Ένας δικηγόρος μου είπε ότι αυτά είναι, γίνονται κατά κρίση. Ε, βεβαίω, ε, κρίση η οποία επηρεάζεται όταν ε, ο πελάτη πληρώνει και μερικά εκατομμύρια δολάρια ω αμοιβή δικηγορική. Λοιπόν, το βασικό πρόβλημα εδώ πέρα με αυτού οι οποίοι διευκολύνουν τους ολιγάρχες είναι ότι πρόκειται για μια πολύ επικερδή εργασία και αυτό είναι και ο σκοπό του βεβαίω και από εκεί πέρα μια επιχείρηση λειτουργεί έτσι ακόμα και σε πολύ ε, περίεργες χώρες όπου θα έπρεπε να είναι πολύ πιο επιφυλακτική. Το αν μπορεί να αλλάξουν αυτά είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε εδώ πέρα να επικεντρώσετε την προσοχή σας ε, και ακριβώς ε, οι διοκτικές αρχές και οι νομοθέτες να δουν λίγο το θέμα της επιβολής των νόμων για το ξέπλυμα χρήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τις εισαγωγικές σας ομιλίες, για την παρουσίαση της κατάστασης, ζωφερής βέβαια. Και βλέπω ότι η συνεδρίασή μας έχει προσελκύσει τον ενδιαφέρον μιας μεγάλης ομάδας ε, μάθητών του Λυκείου Λουτβίχ Φαν Μπέτοβεν της Βόνης. Καλώς ήρθατε. Συζήτηση λοιπόν μεταξύ των βουλευτών μας και των προσκεκλημένων μας. Ακούμε τις ερωτήσεις. Πεντά λεπτά για, την ερω... για τις ερω... απαντήσεις, δηλαδή ένα λεπτό για την ερώτηση και τέσσερα λεπτά για την απάντηση. Παρακαλώ τους συναδέλφους να είναι σύντομοι για να αφήσουμε αρκετό χρόνο απαντήσεως στους προσκεκλημένους μας. Ο κύριος είναι συνεισηγητής από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Πολλές ερωτήσεις έχω. Βέβαια θα περιοριστώ στην πιο, ε, σύντομη, στις πιο σύντομες. Ε, για τον κύριο Ασλοντ και τον κύριο Μπρούξ μας λέτε δηλαδή ότι είστε σε θέση είναι δυνατόν να ε, διαγνωστεί η πορεία, να ανοιχνευτεί η πορεία μέσω τραπεζών αυτών των παράνομων κονδυλίων. Εάν λοιπόν τα ποσά αυτά τώρα έχουν περάσει σε επενδύσεις ή έχουν ε, ρευστοποιηθεί. Τι από τα δύο ισχύει, αυτή είναι η ερώτησή μου. Και επίσης βλέπετε και φοροαπάτες παράλληλα, κάποια άλλες δηλαδή ε, παραβίαση άλλων διατάξεων του νόμου και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει δίωξη για την διακράτηση, την αξιοποίηση τέτοιων ε, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η δεύτερη ερώτηση, κεντρική διαχείριση της ε, εποπτείας για την καταπολέμηση της νομοποίησης παρανομών εσόδων. Ε, αντιλαμβάνομαι βεβαίως τα κίνητρά σας, αλλά ταυτόχρονα αυτό σημαίνει και αυτοψίες από τους αρμοδίους στις διαφορές χώρες και διαρωτώ με εάν οι εποπτικές, τραπεζικές εποπτικές αρχές που ε, και την ε, τραπεζική και την δημοσιονομική σταθερότητα των ε, τραπεζών θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ένα τέτοιο ρόλο ελέγχου της νομοποίησης παρανομών εσόδων. Γιατί εδώ πέρα αυτό θα συνεπαγόταν ε, σύγκρουση συμφερόντων των τραπεζών των ίδιων. Πώς είναι δυνατόν αυτές να ελέγχουν την νομιμότητα των ποσών όταν τα διαχειρίζονται κιόλα. Βέβαια, εδώ πέρα έχουμε κίνδυνο και ως προς την επιβολή των κυρώσεων και ως προς το κύρος ε, και την εικόνα της εποπτείας. Οι υποπτικές αρχές λοιπόν σε ποιο βαθμό μπορούν αυτό να το αναλάβουν και σε ποιο βαθμό θα αρκούσε να αυξηθούν τα πρόστιμα, οι κυρώσεις. Επίσης, τελευταία ερώτηση. Η δέουσα επιμέλεια σε περίπτωση κονδυλίων προερχομένων από τη Ρωσία Πώς μπορεί να υλοποιηθεί, είπε ο κ. Ασλούντ, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε κονδύλια που προέρχονται από την Ρωσία ούτω ή άλλω. Ε, όμως πώς το εννοείται αυτός, πώς είναι δυνατόν αν δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στους χρηματοπιστωτικούς ή άλλους τους θεσμού ε, ή στην πορεία των ε, κονδυλίων. Ποιο είναι το επίπεδο αποδοχή που θα μπορούσαμε να περιμένουμε για του πελάτε, Εάν δεν υπάρχει δηλαδή επαρκής βεβαιότητα και ασφάλεια, τι είδους ε, ε, συναλλαγές μπορούμε να έχουμε με αυτούς τους πελάτες. Ευχαριστώ πολύ για τις τρεις ερωτήσεις, ο κύριος Όσλουντ. Από πού προέρχονται τα κονδύλια και πώς ε, κινήθηκε. Πρώτον, έχει περάσει μέσα από μία αξιόπιστες τράπεζε δεκαετία του 90. Μετά έχει περάσει μέσα από ιδιωτικές αλλά και κρατικές εταιρείες και έχει περάσει και από τη διαδικασία της φόρου αποφυγής. Μην ξεχνάμε ότι όλοι οι Ρώσοι έχουν ε, καταθέσει το εξωτερικό γιατί δεν αισθάνονται ασφαλείς ως κάτοχοι λογαριασμών στη χώρα τους. Και για να περάσω στην τελευταία σας ερώτηση ταυτόχρονα, όταν έχουμε να κάνουμε, όπως είπε ο κύριος Μπρούξ, με αξιωματούχους, κρατικούς υπαλλήλους που δεν είναι δυνατόν να έχουν κερδίσει νόμιμα τα χρήματα αυτά πρέπει να προλάβουμε πριν να δαπανηθούν, γιατί άπαξ και δαπανηθούν δεν είναι εύκολο να τα ανοιχνεύσουμε. Ένα παράδειγμα μπορώ να σας δώσω πριν να ξεσπάσει η τραπεζική κρίση, γιατί ήταν προφανές ότι θα ξεσπούσε λίγο αργότερα, όπως άλλωστε και συνέβη, ε, το 2012 δηλαδή πήγα στην Κύπρο για να ρωτήσω Ρώσοι και Ουκρανοί γιατί να κρατούν τα χρήματα σε αυτές τις τράπεζες και επιχειρήσεις όταν είναι ξεκάθαρο ότι έρχεται κρίση. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι αυτά τα ποσά ανήκαν σε εισαγγελείς, αστυνομικούς, δικαστές και δεν είχαν το δικαίωμα να τα μεταφέρουν σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν δηλαδή τόσο εξόφθαλμα παράτυπη η προέλευση αυτών των εσόδων. Και... Ναι, όχι, λυπούμε. Είναι όμως ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να ανοιχνεύσουμε. Σύντομη απάντηση ας αρχίσει η ανείχνευση από τους αξιωματούχους του δημοσίου. Γιατί εκεί είναι πολύ εύκολο να φανεί. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά ο προλαλή σα έκανε μια σημαντική ε, διάκριση ανάμεσα σε περιπτώσει όπου σαφώ μπορούμε να πούμε ότι είναι παράνομο το χρήμα και σε περιπτώσει όπου δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Όπου επιχειρηματίε έχουν τεράστιε περιουσίε, αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι σαφώ παράνομα τα κεφάλαια αυτά. Οι τράπεζε, οι δικηγόροι και οι λογιστέ ε, θα βρουν αιτιολογικά λόγους για να ελέγξουν αυτά τα λεφτά. Αλλά είναι δύσκολο να γίνει αυτό αμέσω. Και αυτό δείχνει ένα μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει από πίσω. Το να εκθέσουμε το συστημικό πρόβλημα που δημιουργεί αυτήν την κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα πρέπει να έχουμε ε, δυτικές λογιστικές εταιρείες, ας πούμε, μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, που θα λένε τα πάντα. Είναι εντάξει. Ας πούμε, να χρησιμοποιούνται νομίμως κονδύλια των, της Gazprom, ας πούμε, χωρίς να υπάρχουν παραβιάσεις ε, λόγω ενδομιλικών τιμολογήσεων. Έχουμε πρόβλημα να εφαρμόσουμε άμεσα τις κυρώσεις λόγω της νομοθεσίας περί καταπολέμησης της, του του χρήματος. Ε, γι' αυτό δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το λανθάνο, το ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα ε, για την τράπεζα Ντάνσκε. Ξέρουμε από την ε, έκθεση της Επιτροπής Ντάνσκε ότι υπάρχουν τεράστια ποσά ε, που κατά την ε, έρευνα δεν κατάφεραν να εντοπίσουν την προέλευση. Κάποια, ας πούμε, πέρασαν μέσω του Αζερβαϊτζάν ή ξέρουμε, ας πούμε, ότι οι πολιτικοί του Αζερβαϊτζάν ε, ασκούν επιρροή, ας πούμε, στην Ευρώπη. Τις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν ξέρουμε, ας πούμε. Ε, γιατί ακριβώς ε, σχεδιάζονται έτσι, ε, με επαγγελματίες, για να είναι αδιαφανή αυτά τα, τα κανάλια. Ε, και χρειάζονται πολύ προηγμένες ε, έρευνες ε, των διοκτικών αρχών για να τα ανοιχνεύσουμε αυτό. Για την σύγκρουση ανάμεσα στο θέμα της σταθερότητας και της πρόληψης των τραπεζών μπορεί να υπάρξει σύγκρουση εδώ και θα πρέπει οι ρυθμιστικές αρχές που εμπλέκονται σε αυτές τις επιχειρήσεις μπορούν να φοβούνται αν πάρουν δράση, ας πούμε. Ε, από τη μία μπορεί να φοβούνται να πάρουν δράση, ε, να δημιουργήσουν, μπορεί να αρχίσουν να κυκλοφορούν φήμε, α πούμε, και ο κόσμο να θέλει να πάρει τα λεφτά του από τι ή από την άλλη, αν δεν κάνουν τίποτα, α πούμε, να έχουν πρόβλημα με, την, με τον νόμο. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα επίση ε, στο να επιβληθούν μεγάλε κυρώσει. Εγώ Θεωρώ ότι τα πολιτικά θέματα είναι τα πιο σημαντικά που καθορίζουν και τη στάση των τραπεζών. Πέντε λεπτά στον επόμενο μιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Σας ευχαριστώ όλους. Συμφωνώ με όλες τις ε, συστάσεις σας. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω, ίσως ε, πρώτο τον κύριο Μπρούξ, αναφέρατε το ότι ελάχιστοι άνθρωποι έχουν καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος από τους ανθρώπους που τους δίνουν αυτή τη δυνατότητα, λογιστές, τράπεζες κτλ. Πώς θα φροντίσουμε λοιπόν να υπάρχουν επαρκείς κυρώσεις και το βάρος αποδείξεως να αντιστραφεί ώστε να υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για ανθρώπους που κάνουν ε, κάτι τέτοιο και μπλέκονται σε τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες. Αλλιώς, ως δανός δηλαδή, Βλέπω ότι εξακολουθεί να υπάρχει η ατιμορρησία. Δεν κινδυνεύει κανείς να κάνει, όταν κάνει κάτι τέτοιο. Και ε, μετά προς τους κυρίους Όσλοντ και Κίσενμπαουμ υπάρχει αυτή ακριβώς ε, η ανισορροπία μεταξύ του συστήματος που έχουμε δημιουργήσει στην Ευρώπη, ενιαία αγορά, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων κτλ και, με, και των εθνικών αρχών που είναι οι υπεύθυνε ε, για την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας αυτής. Όπως ε, το είπε και η Google, είναι συστημικό το πρόβλημα. Τι μας εμποδίζει στο να γίνει κεντρική αυτή η διαδικασία. Γιατί δεν βλέπω να υπάρχει καθόλου όρεξη για ένα τέτοιο κεντρικό σύστημα καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος ε, χρήματος. Αντιθέτως ε, θα έπρεπε να το θέλουμε γιατί θα δημιουργήσει οικονομική σταθερότητα. Γιατί λοιπόν το πολεμάτος ο πολύ Σας Ευχαριστώ κύριος Μπρούξ. Σας ευχαριστώ. Το ερώτημα για το πώς θα υπάρξει αποτροπή, αυτό νομίζω λέτε, είναι ένα θέμα και πολιτικής βούλησης ε, και δυνατότητας να γίνει κάτι. Νομίζω πως υπάρχει πολιτική σύγκρουση σε πολλές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπερήφανο για το ότι είναι μια χώρα κράτους δικαίου ναι, φήμη τα κτλ. Ε, και όταν ανοίξει αυτό το κουτί της Πανδώρας το υπονομεύουμε αυτό. Και αυτή η εποδός ε, επαναλαμβάνεται τόσο καιρό ώστε είναι τόσο δύσκολο μια κυβέρνηση να δεχτεί ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποιους κλάδους ε, των υπηρεσιών που θεωρεί ότι έχουν τεράστια αξία και παγκόσμια φήμη οπότε ε, είναι κάτι το πολύ μεγάλο μετά και πιο απλή λόγη είναι και πολύ δύσκολο για τις διοκτικές αρχές ε, και χρονοβόρο να ασχοληθούν με τέτοιες υποθέσεις και να τις φέρουν στα δικαστήρια ξέρετε ότι τα εν λόγω άτομα θα επιστρατεύσουν και πολλούς δικηγόρους Οπότε η προσπάθεια αυτή μετά γίνεται τελείως ε, διοικητική και γίνεται και τελείως αχρώμη γιατί δεν υπάρχουν καταδίκες δηλαδή και τα πρόστιμα τα μεγάλα θα είναι για διαδικαστικά ζητήματα αυτό λοιπόν δεν αποτρέπει κανέναν όπως είπατε εσείς ότι πρέπει να γίνει πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσεις να δουν το θέμα της αποτροπής όταν μιλάμε για καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος Θα συμφωνήσω και εγώ ότι οι διώξει είναι πάρα πολύ δύσκολες γιατί θα πρέπει να δείξουν ότι, υπάρχουν, ότι υπάρχει γνώση του αδικήματος και είναι κάπως δύσκολα αυτά να αποδειχθούν. Αλλά ειδικά σε κάποιες μικρότερες χώρες είναι και θέμα δυνατότητας της διοίκησης. Αλλά στις μεγαλύτερες σημαίνει πραγματικά ότι θα πρέπει να αφιερωθούν πολλοί μπορεί να εξοδευτούν πολλά λεφτά και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει. Ο επόμενος πανελίστας ε, ε, έχει επιδείξει μεγάλη δουλειά στον τομέα αυτό. Αλλά είναι, όπως σας είπα, δύσκολο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν κάποιες ε, επιτυχίες τέτοιες περιπτώσεις στους τελευταίους μήνες σε σχέση με τη Βενεζουέλα και τη Μαλισσία αλλά και εκεί πέρα πολύ λίγοι άνθρωποι καταδικάζονται. Όσον αφορά μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία, δεν ξέρω τι το εμποδίζει, δεν έχω ακούσει να υπάρχει πολιτική πίεση από τις τράπεζες. Υποψιάζομαι ότι η δημιουργία μια νέα υπηρεσία βεβαίω αφαιρεί εξουσία από τα κράτη-μέλη και προσθέτει περιπλοκότητα στο σύστημα και θα έλεγα βεβαίως ότι αξίζει να γίνει κάτι τέτοιο αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα διαφοροί συνδυασμοί που θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί από την τωρινή κατάσταση και έτσι θα μπορέσουμε να προσθέσουμε διαφορούς πόρους παραδείγματος χάρη στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, την ΕΣΜΑ δεν χρειάζονται δηλαδή απαραίτητα νέε υπηρεσίε, χρειάζεται μια εντολή πόροι και άνθρωποι και βεβαίω μπορεί να πάει σε έναν ενιαίο υποπτικό μηχανισμό. Γιατί βεβαίω έχουν εκφράσει την επιθυμία να υπάρχει μια προληπτική ε, εποπτεία. Αλλά δεν χρειάζεται άρα να δημιουργήσουμε νέα υπηρεσία οπωσδήποτε. Και η πρόοδος η οποία σημειώνεται μπορεί να είναι μικρή και είναι οπωσδήποτε καλύτερη από το τίποτα. Και υπάρχει ένα χάσμα βέβαιως μεταξύ αυτή τη σταδιακής προσέγγιση και τη ε, ε, προσέγγιση που επιζητεί το μάξιμουμ. Εγώ θα σα έλεγα ακριβώ να βρεθείτε κάπου στην ε, μέση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξαιρετικές παρατηρήσεις. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές τράπεζες κάνουν το αντίθετο γιατί έχουν διαφορετικά κίνητρα στις ΗΠΑ οι τράπεζες την τελευταία δεκαετία έχουν πληρώσει 220 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα. Ξοδεύουν λοιπόν δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για να συμμορφώνονται με την νομοθεσία και θέλουν να μειώσουν αυτό το κόστος. Οπότε τώρα οι αμερικανικές τράπεζες θέλουν ε, οι τελικοί δικαιούχοι να αποκαλύπτονται ε, και να γίνει αυτό μισό της νομοθεσίας. Αυτό το ζητάνε οι τράπεζες, ενώ ε, στην Ευρώπη λένε τι χρειαζόμαστε αυτή τη γραφειοκρατία κτλ. Και λοιπόν αν έτρωγαν περισσότερα πρόστιμα θα έβλεπαν τι το χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ Γκίνερ Χέκμαρκ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ κύριοι για τις παρουσιάσεις αυτές. Απελπισία σε πιάνει, όχι μόνο λόγω των μεγεθών, αλλά και λόγω της απουσίας κατάλληλης ανταπόκρισης και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να κοιτάξουμε κατάματα αυτή την ε, εκθεμελίων απειλή για την ε, Ευρώπη. Πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες από ό,τι βλέπουμε έχουν καταστεί τμήμα αυτού του κυκλώματος και θα ήθελα από εσά να ακούσω πρώτον ποιο είναι το συνολικό μέγεθος. Μιλήσατε για την Εστονική Τράπεζα με 150 δισεκατομμύρια ή κάποια άλλα παραδείγματα που δώσατε, αλλά συνολικά γιατί ποσά μιλάμε. Και δεύτερον, απειλή ως προς την ασφάλεια που μπορεί να φέρουν αυτά τα κονδύλια. Επίση, είπε ο κύριο Όλσον μόλι τώρα ότι οι ευρωπαϊκέ τράπεζε τείνουν την ε, νομοθεσία να την αντιμετωπίζουν μόνο σαν γραφειοκρατική επιβάρυνση. Αλλά δεν θα συμφωνήσω εγώ με αυτό, γιατί αν έχω μια θεία ε, που θέλει να καταθέσει χρήματα ή μια γιαγιά που θέλει να καταθέσει χρήματα ε, σε μια τράπεζα και μπήκε σε τρίτη κατηγορία αποταμίευσης ή εγώ ίδιος 15 χρόνια που είμαι εδώ και που έχω μαζέψει κάποια χρήματα στις Βρυξέλλες ή από τις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να δω λοιπόν, όσο τετριμένο και αν σας φαίνεται, το θεμελιώδες κατά τα άλλα ζήτημα, το πώς το καλό κάτι τέτοιο μπόρεσε να συμβεί με όλη την ομοθεσία που έχουμε. Και για να το προσθέσετε και στις λοιπές απαντήσεις σας, πώς εξασφαλίζουμε την ανείχνευση, την παρακολούθηση και την κύρωση την κατάλληλη σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ λησμόνισα και με συγχωρείτε ο κύριο Χόικ Μαρτίν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Νομίζω ήταν προφανέ, Πρόεδρε, προ του ε, άπαντε. Ναι, α το καταστήσω κι εγώ πιο προφανέ. Ε, ο κύριο Όλσλουν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για να απαντήσω στι δύο πρώτε ερωτήσει. Η εκτίμηση για συνολικό ποσό ρωσικού χρήματος, 800 δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό, χωρίς να ξέρουμε ακριβώ πού και μπορεί να φτάνει και μέχρι 1,3 εκατομμύρια δολάρια το ποσό αυτό. Βέβαια, η νομιμοποίηση παρανομών εσόδων έχει πολύ, πολύ ψηλότερα ποσά, αντιστοιχεί σε πολύ ψηλότερα ποσά, γιατί κυκλοφορεί το χρήμα από την Εστονία και από άλλες χώρες και άρα είναι πολύ ψηλότερα τα ποσά. αν και δεν είναι εύκολο να το κοιτάξουμε. Και βέβαια πολλές φορές τα χρήματα αυτά παρκάρονται στα ακίνητα και βέβαια αποτελούν και απειλή για την ασφάλεια και κάποια από τα χρήματα αυτά μπορεί να ε, μπουν σε κυκλοφορία. Οι κουρανικέ εκλογέ, σε παράδειγμα, τώρα ζωτική σημασία και προβλέπεται ότι μπορούν να κοστίσουν έω και ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ε, από αυτά το, τα 500 εκατομμύρια μάλλον θα τα δώσουν κύκλοι ολιγαρχικών συνδεωμένων με το Κρεμλίνο. Και άρα κατά πάσα πιθανότητα αυτοί που θα εκλεγούν στην Ουκρανία ή μεγάλο ποσοστό αυτών θα έχουν ε, στενή διασύνδεση με τη Ρωσία. Το ίδιο και με την Ελβετία, αν δούμε τα δημοψηφίσματα πόσο μπορεί να κοστίζουν, ε, εάν κοστίζει ένα δημοψήφισμα ε, στη Σουηδία εάν κοστίζουν ε, οι εκλογές ε, κάποια εκατομμύρια δολάρια πόσα μπορεί να είναι από τη Ρωσία και να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Το ίδιο είδαμε με το Brexit και το δημοψήφισμα. Επομένως είναι τεράστια τα ποσά που έχουν φύγει, αλλά ακόμα και μικρό τμήμα αυτών μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση εκλογικών αναμετρήσεων. Ο κύριος Κίρχενπομ, ναι, εκατοντάδες εκατομμύρια ε, μπορεί να νομοποιούνται μέσα από τις τράπεζες ε, αλλά μια γιαγιά ή μια ηλικιωμένη θεία να μην μπορεί να ε, φέρει χρήματα ή να θεωρείται υποπτή αν φέρει χρήματα για να τα καταθέσει στην τράπεζα. Εάν γίνεται λοιπόν τέτοιος έλεγχος για έναν ηλικιωμένο ταξιούχο, δεν υπάρχει λόγος αυτόματα να κινητοποιεί το μηχανισμός ε, διερεύνησης όταν έρχονται μεγάλα ποσά από αλλού. Αλλά εδώ μιλούμε για επαγγελματικά δίκτυα που έχουν εγκαθιδρύσει ε, και υπεράκτιες εταιρείες ε, που η μία συγκαλύπτει την επόμενη. Το είδαμε. Άλλωστε, εκεί όπου είχαμε μικρό αριθμό επιχειρήσεων που μέσα από κάποιους που διευκόλυναν την κίνηση του χρήματος το έφεραν από την κοινοπολιτεία ανεξαρτών κρατών στην Ευρώπη και μπρος πίσω μέσα από αυτές τις ε, ε, επιχειρήσεις ή τις εταιρείε βιτρίνα το είδαμε στην Κτάνης και παραδείγματι είχαν τεράστια ποσοστά ε, ιδιοκτησίας σε αυτήν την εταιρική, στην εστονική εταιρεία και μετά αυτά πέρασαν κατά τρόπο αδιαφανή σε άλλες εταιρείες. Ο έλεγχος μπορεί να γίνεται εάν υπάρχουν και τα κατάλληλα κίνητρα και οι κυρώσεις βεβαίως. Δεν μπορεί κάθε τράπεζα να ελέγχει κάθε εγκληματία, να αποτρέπει την κατάθεση χρημάτων από τον οποιονδήποτε εγκληματία. Από την άλλη όμως δεν είναι και τόσο δύσκολο εκατοντάδες ε, δισεκατομμυρίων δολαρίων ε, σε μια μικρή τράπεζα να μην χτυπήσουν ένα καμπανάκι και να μην ελεγχθούν. Και εδώ έρχομαι και στη σύγκριση με την ε, ηλικιωμένη καταθέτρια. Υπάρχει τρόπος δηλαδή, ο κύριος Μπρούξ. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο στο κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι μια απειλή για την ασφάλεια για να διαφωνήσω με τον κύριο Άσλοντ, ο οποίος μας είπε ότι ε, δεν είναι απειλή ίσως για την ασφάλεια το να μπουν τα χρήματα αυτά σε ακίνητα στο Λονδίνο. Όχι είναι, διότι είναι απειλή για την ασφάλεια το ίδιο το καθεστώς που διατηρείται στην εξουσία χάρη στα ποσά αυτά και στη ε, περιουσία αυτή αυτός που αγόρασε το ακίνητο διεφθαρμένος ή ε, εκτεθειμένος στη δωροδοκία και τη δωροληψία αποτελεί απειλή για τον απλό άνθρωπο στην Ευρώπη. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την απειλή για την ασφάλεια, όχι για το συγκεκριμένη, δηλαδή για το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, για το κάθε νόμισμα που θα πάει, αλλά για το κύκλωμα όλο αυτό και την κυκλοφορία αυτού χρήματος. Επίσης οι μικροκαταθέσεις και πόσο βολικό μπορεί να αξιοποιούνται αυτές. Νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με όλο το σύστημα της ε, συμμόρφωσης των ε, τραπεζών, τραπεζικού τομέα στην νομοθεσία. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε ότι οι διαδικασίες τηρούν την ε, νομοθεσία, δηλαδή δίνουμε την εντολή σε έναν υπάλληλο, σε μια θηγατρική, σε ένα υποκατάστημα καλύτερα να ελέγξει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα και άμα το κάνει θεωρούμε ότι είμαστε ασφαλείς. Πολύ καλά, μπράβο. Και ελέγχουμε έτσι το μικρό καταθέτη. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε μεγάλες καταθέσεις και όταν πρόκειται ο διευθυντής ε, του υποκαταστήματος να ε, δώσει το τυποθήτο για το, την έγκριση για μια κατάθεση, αυτόν τον έχει πείσει κάποιος μεγάλο δικηγόρος, ίσως και με κάποια ποσά. Ευχαριστώ. Για την ε, Danske Bank ε, να σας υπενθυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα θα πάμε στην Εστονία και την Δανία για να ε, συνεχίσουμε τις έρευνες μας. Σας ευχαριστώ κύριε Αγκόμες. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά που ζητήσατε ένα νόμο Μαγνίτσκι για λόγους ξεπλήματος χρήματος. Εγώ το ζητάω από το 2013 για λόγους ανθρωπινών δικαιωμάτων κυρίως, αλλά βεβαίως ε, πολύ σωστά λέτε ότι θα χρησιμεύσει και στο ξέπλυμα χρήματος. Δηλαδή θα σημαίνει στοχευμένες ε, κυρώσεις. Αλλά δεν θεωρείτε ότι οι χρυσές ε, βίζες που εμφανίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και στη ΣΥΠΑ είναι ένας τρόπος να παρακάμψουν τις ε, κυρώσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα η Κομισιόν μετά από πίεση του Κοινοβουλίου έβγαλε μια έκθεση για τις ε, χρυσές ε, θεωρήσεις που είναι πολύ έντονη εκτός από τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Αλλά μία από τις συστάσεις που δεν υπάρχει και θα έπρεπε να υπάρχει είναι πώς ακριβώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ιδέουσα επιμέλεια για τα άτομα που είναι σε καταλόγους κυρώσεων. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Αναφέρατε την περίπτωση Πάξα που ήταν ε, Ένα άτομο το οποίο βγήκε από τις λίστες κυρώσεων στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι υπήρχε ένα ευρωπαϊκό λόμπι για αυτήν ακριβώς τη δουλειά για να βγει ο κύριος Πάξα από τις αμερικανικές κυρώσεις για τον κύριο Κέστενμπαουμ. Συμφωνώ μαζί σας ε, πλήρως και νομίζω αυτό είναι ένα συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρξει να πάει η καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος ε, στην ε, κεντρική εποπτεία των τραπεζών. Έχουν πολλές πορτογαλικές τράπεζες που είναι πλυντηρία για την Αγγόλα. Και και σίγουρα θα υπάρχουν και για τους ε, Ρώσους όπως υπάρχουν ε, ε, για τους Αζέρους κτλ. Λοιπόν αυτές οι περιστρεφόμενες πόρτες, οι μουσικές καρέκλες δηλαδή, μεταξύ δικηγόρων, λογιστών κτλ, συμβούλων, τραπεζών και μετά νομοθετών κτλ. Μήπως αυτό είναι η ουσία του προβλήματος. Τέλος, για τον κύριο Μπρούξ υπουργό ε, εξωτερικών ε, ε, βρίσκεται στην Σιγκαπούρη του Ηνωμένου Βασιλείου και από ό,τι φαίνεται ότι με το Brexit θα γίνει και το Ηνωμένο Βασίλειο ένας φορολογικός παράδεισος. Το συνειδητοποιεί αυτό ο κόσμος. Σας ευχαριστώ κύριο πάμε Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε για τις χρυσές θεωρήσεις και βεβαίως ανέφερα και την περίπτωση Γενάντη Τιμοσέγκο και τον κύριο Ρούτενμπεργκ που είναι και Φιλανδοί πολίτε, δηλαδή πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, δεν μπορούν άρα να μπουν σε κατάλογο κυρώσεων. Απέκτησαν τη δεκαετία του 90 επικότητα σε πιο αθώου καιρού. Αλλά είναι αρκετοί άνθρωποι σε αυτό το καθεστώ και τώρα προσφάτως είδαμε μεγάλο σημαντικό αριθμό πολύ πλούσιων Ρώσων να αγοράζουν υπηκότητα μαλτέζικη και κυπριακή που είναι λόγος για έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των χρυσών θεωρήσεων. Αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι έλεγχοι, είναι ευαίσθητο το ζήτημα και ο Πάσκα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Εξ όσων γνωρίζω έχει χιτήρια αλουμινίου σε 7 ευρωπαϊκές χώρες, Σουηδία, Ιρλανδία και αλλού. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει κάποιος ε, σοβαρός έλεγχος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, γιατί θα πρέπει να δούμε όχι μόνο αυτά τα οποία δεν επιτρέπονται από την σκοπιά της ασφαλείας έχει δίκιο για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπρούξ για το θέμα της εθνικής ασφαλείας αλλά και από την νομική σκοπιά Πολλά εργοστάσια έχουν αγοραστεί στην Ευρώπη, κυρίως στη Βρετανία, αλλά και αλλού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει έναν άλλο τρόπο ελέγχου εθνικής ασφαλείας και νομικού ελέγχου των ξενοπαιδίσεων. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση κάτω δευτερεύων για την περίπτωση Πάσκα βγήκαν από το Αμερικανικό Χρηματιστήριο από τη... λόγω του Αμερικανικού κράτους. Ε... παραμένει όμως ε, προσωπικά ως άτομο στην λίστα των κυρώσεων τώρα για τα ζητήματα του αλουμινίου δεν ε, ξέρω αν μια ευρωπαϊκή χώρα καμία ευρωπαϊκή χώρα έχει ζητήσει κάτι ανάλογο τώρα Ναι, άνε ναι, για τις ε, ανθρώπους αυτούς που διευκολύνουν την κατάσταση και είναι ένα κύκλωμα. Κοιτάξτε, η απειλή που προκύπτει από το να έχουμε μεγάλο χρηματοπιστωτικό κλάδο και μετά εξάρτηση από το ρωσικό χρήμα είναι η πολιτική εξάρτηση πολύ περισσότερο από συγκεκριμένες περιπτώσεις ή παρεμβάσεις και το θέμα πηγαίνει πέρα από τις τράπεζες. Είναι ευρύτερο το ζήτημα και περιλαμβάνει και τους διαχειριστές κεφαλαίων, λογιστές, δικηγόρους και τους ε, υπόλοιπους. Τώρα, για την αποτελεσματικότερη υποπτία. Αυτό είναι πρόβλημα παντού, ειδικά εκεί όπου είναι υπερμεγέθης ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Υπάρχει θέμα επιρροής και όλοι όσοι παρέχουν επαγγελματικέ υπηρεσίε είναι μέρος ε, του φαινομένου. Αυτό το οποίο είπατε για τις πορτογαλικές τράπεζες και την Αγγόλα είναι ενδιαφέρον γιατί το μπορεί να, τι, μπορεί να γίνει καλύτερα με το υφιστάμενο πλαίσιο. Όπως λέτε οι πορτογαλικές τράπεζες εμπλέκονται σε δραστηριότητε ε, στην Αγγόλα. Δεν ξέρω πώ ε, έχουν αλλάξει τα πράγματα με τη νέα κυβέρνηση στην Αγγόλα και το καθεστώ Ντο Σάντο. Αλλά τουλάχιστον δύο πορτογαλικές τράπεζες αγοράστηκαν την Ιζαμπέλ Ντοσάντος και ξεκίνησε τελικά η Ευρωπαϊκή Αρχή η διαδικασία κατά των πορτογαλικών εποπτικών αρχών και έκρινε ότι παραβιάστηκε το ευρωπαϊκό δίκαιο. δεν θυμάμαι ακριβώς την σειρά, αλλά πρώτα οι πορτογαλικές αρχές και μετά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να δουν την αλλαγή αυτή της ε, ιδιοκτησίας. Οπότε μπορεί να είναι μια χαρά οι νόμοι στα χαρτιά και να του έχουμε σχεδιάσει μια χαρά, αλλά αυτό το οποίο μετράει είναι η επιβολή. Οπότε σαφώς εδώ πέρα υπήρχαν κανόνες που θα μπορούσαν να καλύψουν ε, πολιτικά πρόσωπα σε μια πολύ διεφθαρμένη χώρα. Κι όμως αυτό συνέβη με τις πορτογαλικές τράπεζες και δεν είναι πολύ δύσκολο όμως να το αποτρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ γρήγορα για το, για το Λονδίνο που θα γίνει Σιγκαπούρη μετά το Brexit. Είναι πραγματική απειλή. Το έχει πει και η Τερέζα Μέη, ε, το έχουν πει και άλλοι Βρετανοί πολιτικοί. Ε, το Foreign Office και η κυβέρνηση προστατεύει τα υπερπόντια εδάφη τα οποία λειτουργούν ως φορολογική παράδειση και συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά το Brexit νομίζω ότι είναι πιθανό ό,τι και να γίνει η, το, η δυνατότητα του, του να ασκεί λόμπι το City να γίνει ε, ακόμα πιο έντονη. Ήδη είναι πολύ ισχυρή ε, και θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή και αυτό που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η χρηματοδότηση ας πούμε και οι κανόνες που ισχύουν στα offshore ε, θέλουν μεγαλύτερη ακόμη χαλάρωση των κανόνων. Η απουσία της ε, Βρετανίας από την Ευρώπη θα σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν θα φοβάται ε, το αν θα ακουστεί ή όχι η φωνή της στην Ευρώπη. Αυτό που θέλει, θα θέλει θα είναι προστατεύσει τα υπερπόντια εδάφη ε, και μπορεί να προσπαθήσει να κάνει μια αντιστάθμιση διευκολύνοντας τα πράγματα για, τους, για τα offshore. Και αν υπάρχουν απειλές, μια και θα είμαστε και εκτός της Ευρώπης, ε, υπάρχει κίνδυνος πραγματικά να κινηθούμε προς πολύ επικίνδυνα νερά, ας πούμε, και να γίνουμε ένα είδος Παναμά, ας πούμε, κάτι που θα είναι μεγάλη απειλή για όλους. Θα μιλήσω ισπανικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις ομιλητές. Τα είπατε όλα. Πήρατε σοβαρές θέσεις, κάνατε σοβαρότατη ανάλυση, κάνατε πολύ ωραίες συστάσεις και μιλήσατε για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια δομή κινήτρων για να αποτρέψουμε τους τεράστιους αυτούς κινδύνους. Γιατί μιλάμε για κλεπτοκράτες από τρίτες χώρες ε, οι οποίοι ε, φέρνουν τη διαφθορά στις χώρες μας σε πολύ σημαντικούς τομείς. Και επιπλέον υπάρχει και εκλογική απειλή, γιατί όταν οι κλεπτοκράτες έχουν γεωστρατηγικές, συμφέροντα, τότε εμείς έχουμε, αντιμετωπίζουμε τεράστιους κινδύνους. Οι δημοκρατίες μας αντιμετωπίζουν τεράστιους κινδύνους. Είπατε ότι θα πρέπει να μεγεθυνθεί ε, η αποτροπή θα πρέπει να έχουμε αρκετό προσωπικό, αρμόδιο προσωπικό, ε, με τα κατάλληλα ε, με τις κατάλληλες δεξιότητες, ούτω ώστε να διώκονται τα, όλα αυτά τα εγκλήματα όπως η φυγή κεφαλαίων και άλλα συναφή εγκλήματα. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε τα τελευταία χρόνια είναι να προστατεύσουμε τις πηγές μας, τους καταγγέλλοντες, ε, αυτούς που καταδίδουν ε, τις παράνομες ε, προβληματικές δραστηριότητες οι οποίες συμβαίνουν και που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να ανοιχνευτούν. Ξέρουμε μέχρι στιγμής ότι όλοι, προσπάθησαν, όλοι όσοι προσπάθησαν να αποκαλύψουν τέτοια αδικήματα είχαν κακό τέλος. Έτσι, ακούσαμε εμπειρίες και μαρτυρίες και εδώ, στο Κοινοβούλιο, και ξέρουμε τι έχει συμβεί σε πολλούς από αυτούς τους καταγγέλλοντες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Πέρα από την προσπάθεια εφαρμογής των συστάσεων που μας είπατε, πιστεύετε ότι μια κωδικοποίηση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ούτω ώστε για αποδεδειγμένα εγκλήματα, για συγκεκριμένες ποσότητες χρήματος, ε, να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να καταγγέλουν αυτά τα αδικήματα. Για να σταματήσουμε τόσες πολλές ε, δραστηριότητες ξεπλήματος χρήματος και μάλιστα δισεκατομμυρίων ε, ευρώ. Και φυσικά να σταματήσουμε και τα, και τα συναφή εγκλήματα και αδικήματα. Κύριο Σάσλου, ευχαριστώ. Σωστά αυτά που είπατε για την κλεπτοκρατία. Αλλά η ε, διαφθορά είναι μέσω υβριδικού πολέμου. Αγοράζεις, εξαγοράζεις πολιτικούς. Οι Ρώσοι δεν αγοράζουν κόμματα, δεν αγοράζουν χώρες, αγοράζουν πολιτικούς. Και το κάνουν σε διαφορετικά κόμματα. Είναι ένα πολύ φθηνό, έξυπνος, οικονόμος τρόπος για να ασκήσεις επιρροή. Και αυτό ε, απαιτεί πολύ αυστηρούς κανόνες ε, διαφάνειας και για το λόμπι και για τους ίδιους τους πολιτικούς οι οποίοι θα πρέπει να αποκαλύπτουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Έχετε, έχει γίνει σε κάποιες χώρες, ε, αυτό το, υπάρχει αυτό το πλαίσιο, αλλά δεν γίνεται παντού. Ένα άλλο κίνητρο είναι ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν το δικαστικό σύστημα δικαστικές αρχές ε, της Ρωσίας ζητούν από διάφορες χώρες να δεχτούν τις ρωσικές δικαστικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά τις ε, κόκκινες προειδοποιήσεις ε, που αφορούσαν συλλήψεις. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει συλληφθεί 7 φορές λόγω του ότι υπάρχουν αυτές οι κόκκινες ειδοποίησεις των Ρώσων. Ζητάνε από τις ΗΠΑ τη λεγόμενη αποκάλυψη πληροφοριών και ζητούν και την πτώχευση και κανονισμούς πτώχευσης να εφαρμοστούν. Διάφορες, εν πάση αποφάσεις των ρωσικών δικαστηρίων που θέλουν να γίνουν σεβαστές. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανασκευάσει ε, τις αποφάσεις πολλών ε, ρωσικών φορέων, γιατί οι αποφάσεις τους δεν βασίζονται στο κράτος δικαίου. Υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα στην Κύπρο. Αλλά όχι μόνο στην Κύπρο. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Στο πρώτο τμήμα της ομιλίας σας είπατε ότι υπάρχει διαφθορά ε, στο χρηματοπιστωτικό τομέα και εκλογική ε, απειλή. Ε, σίγουρα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δημιουργείται εκλογική απειλή και ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση ενός ε, πα, ε, δανείου από μια ρωσική τράπεζα σε μια εταιρεία. Πρόσφατα έγινε μια μελέτη για αυτό το θέμα και υπήρχαν δύο ενδιαφέροντα στοιχεία. Η τράπεζα που όπου ο Ρώσος ε, αξιωματούχος ας πούμε ζήτησε να ελέγξει αυτό το αίτημα ε, σε μία, σε μία, ε, το έδωσε αυτό το δάνειο, ήθελε να το δώσει μάλλον σε μία εταιρεία πλασματική. Στην πραγματικότητα ήταν ένα σχήμα αυτό που είχε κανονιστεί στη Ρωσία και όταν διαλύθηκε η τράπεζα, ε, το δάνειο αυτό είχε πάει στην πλασματική εταιρεία και μετά είχε πάει σε μια βιομηχανία που είχε πάρα πολλές συμβάσεις σε διάφορες χώρες ε, και με το Υπουργείο Άμυνας της Συρίας ε, και υπήρχαν εδώ λοιπόν και βρέθηκαν σχέσεις ανάμεσα στην Συρία, το Υπουργείο Άμυνας και τον Ρωσικό στρατό. Τώρα, για του ε, καταγγέλλοντε. Ο συνάδελφο μπορεί να μιλήσει καλύτερα, ο κ. Μπρούξ μπορεί να μιλήσει καλύτερα για αυτό το θέμα. Ε, το να προστατεύουμε του καταγγέλλοντε και να ενθαρρύνουμε αυτού που έχουν πληροφορίε να τι αποκαλύψουν θα αυξήσει τον αριθμό των υποθέσεων που φτάνουν στο κοινό και στου αρμοδίου. Ε, επίσης όμως ε, θα έχουμε και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία στη διάθεσή μα. Αλλά ακόμα και πολλά αποδεικτικά στοιχεία θα είναι πολύ δύσκολο. Παραδείγματο χάρη πρόσφατα στην Ισπανία ε, έγινε μια δίωξη εναντίον ε, κάποιων που κάνανε ξέπλυμα ε, ρωσικού χρήματος. Αλλά ήταν δύσκολο να φτάσουν σε καταδικαστική απόφαση. Και θα είναι δύσκολο και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για το θέμα των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, whistleblowers. Ε, με ελάχιστε εξαιρεσει η ζωή του έχει καταστραφεί από την καταγγελία ε, είτε βρέθηκαν άνεργοι είτε η προσωπική του ε, ζωή έχει διαλυθεί αυτό πρέπει να έχετε υπόψη λοιπόν ότι πρέπει να προσφέρετε ισχυρά κίνητρα αντίστροφα δηλαδή με την έννοια της ανταμοιβή όπως υπάρχει στις ΗΠΑ για να ε, καταγγείλει κάποιος ένα δίκημα. Ο Μπράντον Μπέκερφελντ είναι η πιο γνωστή περίπτωση ε, μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος στις Πολιτείες Κατήγγειλε ε, φόρο διαφυγή εκτεταμένη στη UBS που δεν θα είχε διερευνηθεί αν δεν υπήρχαν οι καταγγελίες, όπως και πολλά άλλα εγκλήματα. Αυτό πρέπει να κάνει λοιπόν η Ευρώπη. Ένα πρόβλημα βέβαια είναι στην νομοποίηση των παρανόμων εσόδων ότι οι οργανισμοί οι οποίοι θα ε, φυλάξουν τα χρήματα αυτά, τα προϊόντα παράνομων ε, δραστηριοτήτων, δεν είναι ευαισθητοποιημένοι ώστε να καταγγέλουν. Και βέβαια αν κάποιος από τη Ρωσία κάνει μια τέτοια καταγγελία, δεν πρόκειται να τον ανταμείψει στο Κρεμλίνο. Κάποιο άλλο τύπου κίνητρα πρέπει να βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπωσδήποτε όμω θα έξω το κόπο να διερευνηθεί μια τέτοια δυνατότητα. Ο κύριο Γκίγκολτ Πράσινη. Ευχαριστώ πολύ. Ένα θέμα που κάποιοι από σας ανέφεραν, αλλά δεν συστήσαμε διεξοδικά σε μια σειρά από ειδικέ επιτροπές, είναι ο ρόλος της Κύπρου στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του, αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά την ροή παράνομων εσόδων βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη και την ε, διοχέτευσή του σε άλλα σημεία του κόσμου. Εσείς κύριε Κύρχη έχετε κάνει σχετικές δημοσιεύσεις στο παρελθόν. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την παρουσία ρωσικού χρήματος στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα και κυρίως σε σχέση με την ε, δομή της ιδιοκτησίας αυτού του χρήματος και επίσης και οι τρεις σας μπορείτε να μας πείτε μια εκτίμηση για το πόσο σοβαρή είναι η εμπλοκή των ε, αρχών στην Κύπρο προς την υλοποίηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση παράνομων εσόδων. Τι γνωρίζετε, κύριος Κύρχιπαουμ. Κύρχενμπαουμ. Ναι, για την ε, πρώτη ε, ερώτηση και την παρουσία ρωσικού χρήματο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τη Κύπρου. Έχει ιστορικά σημαντικέ διαστάσει. Ο διοικητή τη Τράπεζα τη Κύπρου, ύστερα από μια σειρά γεγονότων και σκανδάλων που αναδύθηκαν στι ΗΠΑ, που αποκαλύφθηκαν στι ΗΠΑ και αφορούσαν και την Κύπρο, έκανε σχετικέ δηλώσει και ε, ανήγγειλε κυρώσει σε σχέση με τον έλεγχο και των καταθέσεων στην Κύπρο. Με συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία όμως δεν νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικά, γιατί τα ποσά των καταθέσεων δεν αναφέρονται σε ένα συλλογικό επίπεδο ιδιοκτησίας. Δηλαδή, αποκαλύπτει τον αριθμό του λογαριασμού με το όνομα εκείνου που έχει δηλώσει πως έχει ρωσική υπηκότητα ή της εταιρεία ενδεχομένω με έδρα η καταστατική η λειτουργική στη Ρωσία. Αλλά αυτό δεν μας λέει πόσα από τα χρήματα αυτά έχουν περάσει από ρωσικές εταιρείες ή σε άλλες εταιρείες μέσα εταιρείε ή σε άλλε εταιρείε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σε αλλες εταιρειε επί παραδείγματι, τράπεζα της Κύπρου, όταν κατέρευσε και το Μπέιλινγκ που της προσέφερε η Τράπεζα της Κύπρου, πολύ σημαντικό, οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη Ουκρανών και Ρώσων ολιγαρχών που είχαν τις μεγαλύτερες καταθέσεις να έχουν και την πλειοψηφία στο, του μετοχικού κεφαλαίου και άρα στη συνέλευση των μετόχων. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε και μιλώ για κυπριακά δεδομένα ε, δύο-τρεις μεγάλες εταιρείε, 50% έχει η Τράπεζα της Κύπρου, η ελληνική που έχει γίνει κυρίως διαχείριση επιχειρηματικών ε, κεφαλαίων και η ICB που διαχειρίζεται ρωσικά κεφάλαια, αλλά και κάποιες μικρότερες, η Αναπτυξιακή Τράπεζα Κύπρου και άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες που είναι παρούσες εκεί. Πάντως αυτό που βλέπουμε είναι πολύ έντονη παρουσία υπηκών της ε, κοινοπολιτείας ανεξαρτητών κρατών ήρω της Ρωσίας, ειδικότερα στο μετοχικό κεφάλαιο. Τσαϊκόφσκι παραδείγματι που μετά ανέλαβε ο Τσέρεβεμπερκ με παρουσία στα διοικητικά συμβούλια και το μετοχικό κεφάλαιο. Μάλιστα αυτός έχει υποστεί σημαντικέ ε, κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Όμως φαίνεται ακόμα να επηρεάζει το ε, μετοχικό κεφάλαιο ε, κυπριακών τραπεζών. Η ελληνική, επί παραδείγματι, ε, έχει ένα μεγάλο μέτοχο που είναι εταιρεία λευκορωσική ηλεκτρονικού τζόγου με ρίζες και στην κοινοπολιτεία και τη Ρωσία και γενικά υπάρχει μια ομικλώδης κατάσταση και η τρίτη, η RCB ρωσική τράπεζα, το λέει και το όνομά τη. Η VTB έχει το μεγαλύτερο ποσοστό των μετοχών της, ρωσική τράπεζα. Η Ακρίτσια την ε, αγόρασε σε ένα βαθμό και όταν αυτή κατέρευσε πέρσι, ο Ζημάριν, διευθύνων σύμβουλος, ακόμη, αγόρασε μεγάλο πακέτο μετοχών και ανακοίνωσε σε κυπριακό μέσο ότι ε, η χρηματοδότησή του προερχόταν από την RCB σε μεγάλο βαθμό. Άρα και εκεί ήδη γεννήθηκαν ερωτήματα για το από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά και πώ έγιναν συναλλαγέ. Επομένω, οι τρει μεγάλε τράπεζε ε, τη Κύπρου έχουν διασυνδέσει με την ε, Ρωσία και την κοινοπολιτεία και βλέπουμε και διαπλοκή και πολιτική επιρροή. Μεγάλη εξάρτηση όπως και να έχει υπάρχει στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου γενικά και στις ε, ε επαγγελματικέ ή χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δηλαδή διαχείριση μετοχικών πακέτων, επενδύσεις, δικηγόροι και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι σαφής η παρουσία τους εκεί. Κύριο Όσλον, ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ εξαιρετική η απάντηση του κύριου Κίρχενμπαου, αλλά θα προσθέσω ένα-δύο πράγματα κι εγώ. Το 2013 έγινε διάσωση τραπεζών με την κρίση που ήταν όλο βρώμικο χρήμα, γιατί το καθαρό χρήμα είχε ήδη φύγει και είχε υπάρξει μια περίοδος προειδοποίησης, καθώς η κατάρρευση των τραπεζών προήλθε από τα ελληνικά ομόλογα το, το Μάρτιο του 2015 με την πάυση πληρωμών και 12 ε, συγγνώμη και με την πάυση των πληρωμών και ε, αυτό οδήγησε στην κρίση στην Κύπρο. Άρα όλοι όσοι είχαν καθαρό χρήμα πρόλαβαν να το αποσύρουν. Το Διεθνές Νοσματικό Ταμείο το 2013 έκανε μια έρευνα εγκληματολογικού χαρακτήρα της παρουσίας ρωσικού χρήματος στην Κύπρο και κατέληξε στην παρουσία 36 εκατομμυρίων δολαρίων εκεί. Σημαντικά ποσά. Μόνο 14 όμως δισεκατομμύρια από τα ποσά αυτά είχαν πράγματι επενδυθεί στην ίδια την Κύπρο. Άρα ήταν πολύ μικρότερο το ποσό που ήταν εκεί επενδυμένο. 70.000 Ρώσοι υπηκόοι ζουν στην Κύπρο. Μπορεί να έχουν εντωμεταξύ περισσότεροι από αυτούς ήδη πάρει και ε, την υπηκότητα την Κυπριακή. Στη Λεμεσό όποιος πάει θα δει ότι οι, τα πόστερ, οι αφήσει στους δρόμους, οι πινακίδες είναι στα ρωσικά. Πολλές από αυτές τις πινακίδες ε, ε, απευθύνονται σε Ρώσους ταξιούχους για την αγορά κινήτων αν έχουν βαρεθεί το κρύο και θέλουν να ζήσουν στον ήλιο. Ε, χρειάζεται λοιπόν μεγάλο ξεκαθάρισμα. Και τώρα φαίνεται ότι απαιτείται η πλήρης και διεξοδική αναφορά του τελικού δικαιουχούμε βάσει τι τελευταίε οδηγίε οδηγίες 4η και 5η για την νομοποίηση παρανόμων εσόδων στην Κύπρο. Φαίνεται τουλάχιστον να, συμμο... τουλάχιστον να συμμορφώνονται με αυτήν, αλλά ταυτόχρονα μα λένε οι αρχέ ότι έχουν κλείσει 15.000 τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς δεν ήταν δυνατό να διαγνωστεί η προέλευση των ποσών που ήταν εκεί στους λογαριασμούς αυτούς. Άρα γίνεται αρκετή δουλειά η RCB που ανέφερε ο Τζόσουα Βίρχενμπαουμ. Τη βλέπουμε στα Panama Papers. Έδωσε 650 ε, εκατομμύρια δολάρια ε, δάνειο στον Ρολντούκιν, τον τσελίστα φίλο του Πούτιν, η RCB, που δεν φαινόταν πουθενά. και υπάρχει μια κυκλική ροή χρήματο που φαίνεται να θέλησε να συγκαλύψει αυτό το δάνειο που θα ήταν χωρίς βέβαια ε, επιστροφή, χωρίς ε, ε, αποπληρωμή και έγινε μια κυκλική ροή χρήματο για να καλυφθεί αυτό το χαμένο χρήμα. Άρα υπάρχει εμπλοκή, τουλάχιστον τη RCB. Κύριος Μπάι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σταθούμε στην περίπτωση του Μουκτάρα Μπλιέζοφ Καζάκου, υπηκόου, ο οποίος ε, ισχυρίζεται πως ε, η Μόσχα και η Αστάνα τον διώκουν συντονισμένα ενώ έχει καταδικαστεί στη χώρα του για υπεξαίρεση 6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2005 έως το 2009 ως διοικητής της BTA της Καζακικής Τράπεζας. 6 δις δολαρίων. Πρώτα λοιπόν ε, φυγαδεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές μετά από τις Γαλλικές βάση εντάλματος διεθνούς από το Καζακστάν, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Το 2012 το δικαστήριο του Αγγλικό επιβεβαίωσε μια καταδίκη για 4 δις δολάρια και μετά στις διαδικασίες αυτές τις δικαστικές προσπάθησε αυτός ο κύριος να ε, εξαπατήσει και τις δικαστικές αρχές της Βρετανίας παρουσιάζοντας πλαστά έγγραφα και έτσι καταδικάστηκε από τις δικαστικές αρχές για προσβολή της δικαιοσύνης σε 22 μήνες φυλάκιση. Όμως φυγαδεύτηκε στην Γαλλία 29 Δεκεμβρίου του 2016 μήνες μετά την υπογραφή από τον Υπουργό ενός ε, εντάλματος ε, ε, έκδοση σταμάτησαν οι διαδικασίες εις βάρος του παρά την απόρριψη της νιωστής προσφυγής του στη δικαιοσύνη είναι σε επίπεδο ακυρωτικού. Και συνεχίζεται αυτή η περιπέτεια στο Καζακστάν, όπου οι αρχές ε, τον υποπτεύονται πως έδωσε και την παραγγελία για την δολοφονία του κυρίου Τάτη τότε προέδρου της τράπεζας Τζάναλεμ το 2004 δολοφονήθηκε της τράπεζας που μετά ονομάστηκε BTA και έτσι βρέθηκε ο κύριος Ασλιεζόφ ως πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου της εν λόγω τράπεζας. Ο κύριος Ασλιεζόφ λοιπόν κατά τη διάρκεια της αυτεξορίας του ίδρυσε και μια τράπεζα με το όνομα Open Dialogue ε, με πολύ σημαντικές επενδύσεις σε κεφάλαια από ό,τι φαίνεται από διάφορες περιοχές ε, ύποπτη για διάφορες δραστηριότητες ε, που φαίνεται πως συναγωνίζεται και τις δραστηριότητες του κυρίου Σόρος. Ερωτώ λοιπόν, ξέρουν οι ομιλητές μας που βρίσκεται ο κύριος Αμπλιέζοφ, εάν βρίσκεται στη Γαλλία θεωρείται ε, σωστό να μπορεί στην πατρίδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με όλες του τις καταδίκες να κυκλοφορεί ελεύθερος και ανενόχλητος. Δεύτερον, έχετε εσείς κάνει έρευνα για αυτά τα δισεκατομμύρια δολάρια που έγιναν Αέρα ε, αέρας και αν, ε, να, αν όχι πρόκειται να κάνετε τη σχετική έρευνα και τρίτον πρόεδρε εσεί σκοπεύετε ως πρόεδρο πρόεδρος της 3 να ζητήσετε ειδική ακρόαση για την υπόθεση Αμπλιαζόφ που έχει πάρει τέτοιε διαστάσεις εντωμεταξύ ή απλώ αρκεί να καταγγέλλετε τη Ρωσία να δηλώνετε εχθρή του Βλαντιμίρ Πούτιν ή, της, ε, ή του Καζακστάν του Ναρζεμπαϊλεφ για να θεωρήσετε να θεωρείτε ότι έχετε περάσει την κολυμβήθρα του Σιλοάμ για κάθε παράτυπο πράξη. Η συστηματική απαγγελία ισχυρισμών και κατηγοριών εις βάρος της Ρωσίας δεν απαλλάσσει κανέναν άλλον από τα θύματα ή αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι θύματα. Σα ευχαριστώ να απαντήσω στην τελευταία ερώτηση για μια πιθανή ακρόαση. Η ακρόαση ξέρετε ότι απαιτεί τη συμφωνία των συντονιστών, των πολιτικών ομάδων και τη διάσκεψης των Προέδρων, αλλά πλησιάζουμε στο τέλος της εντολής, οπότε ε, δεν υπάρχει δυνατότητα νομίζω. Θέλει κάποιο να σχολιάσει κάποια από τι ερωτήσεις. Κύριο Κίσενμπαουμ, δεν ε, γνωρίζω την περίπτωση αυτήν και το ότι κάποιος μπορεί να κλέβει στη Ρωσία και μετά να λέει ότι είναι θύμα διώξεων, ε, οπωσδήποτε μπορεί να ισχύει. Αλλά τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν την ξέρω. Εσείς, να εγνωρίζω ναι, γνωρίζω την περίπτωση και το βρίσκω λίγο δύσκολο να κρίνω και δεν το κάνω. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το κομμάτι της συνεδρίασής μας. Ευχαριστώ πολύ τους καλεσμένους μας. Είμαι σίγουρος ότι λάβαμε πολύ σημαντικές ε, πληροφορίες. Να σας ευχαριστήσω. Κάνουμε μια διακοπή τριών λεπτών και θα συνεχίσουμε με το επόμενο πάνελ. Well, dear colleagues, let's, let us get ready for another panel of Tech 3 Committee. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο επόμενο πάνελ. Let us start the second panel, which is on the specific... Να με λοιπόν στο συγκεκριμένο πάνελ για την υπόθεση Μαγνίτσκι. Καλώς ορίζω τους ομιλητές μας, τον κύριο Μπιλ Πράντεπ, συνειδητής ε, και διευθύνων σύμβουλος ε, της εταιρείας Hermitage Capital Management, ένα επενδυτικό ταμείο το οποίο κάποια στιγμή ήταν ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Ρωσία, χαρτοφυλακίου και μετά από δραστηριότητα 10 ετών στην ε, Ρωσία του αρνήθηκαν να μπει στη χώρα το 2005 ως ε, απειλή για την εθνική ασφάλεια. Μετά τον θάνατο στην φυλακή το 2009 του Σεργέη Μαγνίτσκι, Ρώσου δικηγόρου και ελεγκτή που εκπροσωπούσε την εταιρεία του κυρίου Μπράουντελ, ο κύριος Μπράουντελ ε, ζήτησε από το Αμερικανικό Κογκρέσο να περάσει τον λεγόμενο νόμο Μαγνίτσκι για τις ρωσικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον οποίον τελικά υπέγραψε ο πρόεδρος Ομπάμα το 2012. Καλώς ορίζω και τον κύριο Ιντεσίμα, ο οποίος είναι επικεφαλής της Γραμματείας Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος είναι επικεφαλής της ε, έκθεσης ε, Μαγνίτσκι και λοιπόν που συζητήθηκε στην ε, κοινοβουλευτική διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 22 του μηνός. Καλώς ήρθατε. Ο καθομιλητής θα έχει χρόνο να κάνει την εισαγωγή του, τις αρχές του παρατηρήσεις και ο κ. Πράτολ έχει προετοιμάσει μια εισαγωγή 10 λεπτών. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τον χρόνο και ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε για να πω αυτήν την ιστορία. Θα σας πω την ιστορία της πτυχής ξεπλήματος χρήματος ε, του Μαγνίτσκι. Έχω και μια παρουσίαση PowerPoint και θα ήθελα να κοιτάξετε τις οθόνες ε, και ελπίζω να μιλήσω αρκετά γρήγορα για να τα πω όλα. Η περίπτωση Μαγνίτσκι ξεκίνησε το 2007 όταν διεπράχθη ένα μεγάλο οικονομικό έγκλημα. 230 εκατομμύρια δολάρια φόρων που είχε πληρώσει η εταιρεία μου στο ρωσικό κράτος ε, κλάπησαν από το ρωσικό κράτος, από κάποιους αξιωματούχους. Ο Μαγνίτσκι, ο δικηγόρος μου, ε, ερεύνησε το έγκλημα και κατέθεσε κατά των αξιωματούχων και σε αντίπεινα συνελήφθη, βασανίστηκε επί 358 ημέρες και τελικά δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2009, 37 ετών. Μετά τον θάνατό του, ξεκίνησα μια εκστρατεία για να δικαιωθεί ο Σιγκέ Μαγνίτσκι με δύο σκέλη. Υπήρχε το πολιτικό σκέλος όπου ε, προσπαθούμε να περάσουμε τον σχετικό νόμο και το ποινικό σκέλος. Το ποινικό σκέλος ερώτησε ένα, έκανε ένα πολύ απλό ερώτημα. Ποιος πήρε τα λεφτά, τα 230 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό ε, θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε και υπάρχουν ε, νομίζω κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα που βγάλαμε από την έρευνα αυτή. Το πρώτο στοιχείο στην έρευνα για όσον αφορά το ποιος πήρε τα λεφτά ε, ήταν, ε, ήρθε από κάποιον άνθρωπο ονόματι Αλεξάνδρ Περτσπελίτσκι, ο οποίος ανήκε σε μια ε, εγκληματική οργάνωση, τσακώθηκε με τους υπόλοιπους και ήρθε και μας έδωσε πληροφορίες. Οι πληροφορίες μας έδωσε ήταν το εξής. Ήταν το άτομο εντός του ρωσικού κράτους που ήταν υπεύθυνο για την παράνομη αυτή επιστροφή φόρου των 230 εκατομμύριων. Ήταν η κυρία Όλγα Στεπάνοβα, Κάποια από αυτά τα λεφτά, 11,7 εκατομμύρια, είχαν πάει στον, στο όνομα του συζύγου της στην Credit Suisse. Μας έφερε τα έγγραφα. Διαβάσαμε τις πληροφορίες στον Ελβετό Ισαγγελέα, ο οποίος πάγωσε τα χρήματα. Κατόπιν, ο Αλεξάνδερ Πρεπλίτσνη επίσης ε, απεβίωσε σε ηλικία 44 ετών, ενώ δεν είχε άλλα προβλήματα υγείας στο παρελθόν, στο σπίτι του στο Σάρι. Η αστυνομία δεν ερεύνησε περαιτέρω την υπόθεση. Το 2012 λάβαμε και άλλες ε, πληροφορίες για το έγκλημα αυτό, για τα 230 εκατομμύρια, δηλαδή το που κατέληξαν εντός των ρωσικών τραπεζών και πώς έφυγαν εκτός των ρωσικών τραπεζών και πήγαν στη Μολδαβία. Νομίζαμε ότι είχαμε κάνει μεγάλη ανακάλυψη, αλλά μόνο μέχρι τη Μολδαβία είχαμε φτάσει. Τελικά όμως ε, είδαμε και άλλα πράγματα όταν ε, μια ΜΚΟ για το οργανωμένο έγκλημα κατάφερε να βρει τον φάκελο μιας ε, Μολδαβικής τράπεζας ονόματι Banco de Economy που έδειξε ότι τα λεφτά πήγανε σε Μολδαβία, ε, Εστονία, Λιθουανία, Λετονία Και υποβάλαμε τις σχετικές ε, πληροφορίες, σχετικές χώρες και ξεκίνησαν εκεί ποινικέ υποθέσεις. Το επόμενο μεγάλο βήμα και επιτυχία μας ήταν από το περιοδικό Barons και το OCCRP που ανακάλυψαν ότι κάποια από αυτά τα λεφτά κατέληξαν στη Νέα Υόρκη. Και από αυτές τις ε, πληροφορίες ζητήσαμε από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει μια έρευνα. Πάγωσαν αρκετά ε, κονδυλία και ανακάλυψαν ε, ότι τελικά κάποια από αυτά πήγαν στον κύριο Ντένις Κάτσιβ, γιο του Πιότρ Κάτσιβ, ε, υψηλό βαθμό αξιωματούχου και τελικά συμβάστηκαν με το Υπουργείο Δικαιοσύνη με ένα πρόστιμο 6 εκατομμυρίων. Στην Ελβετία δεν ήταν τόσο τυχεροί και στην Ολλανδία, όπου επίσης έχουν παγώσει τα λεφτά τους. Βρήκαμε 7,8 εκατομμύρια δολάρια που ανήκουν στην οικογένεια Κατσίβ στην ε, Ελβετία και 3 εκατομμύρια ευρώ των ιδίων στην Ολλανδία. Έχουν παγώσει οι λογαριασμοί αυτοί και στις δύο χώρες και κρεμούν οι ποινικέ υποθέσει. Επίση από την έρευνα στην Εστονία, βρήκαμε και αρκετά χρήματα να πηγαίνουν στην Γαλλία. 28 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 28 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησαν οι Γάλλοι εισαγγελεί σε μια έρευνα, πάγωσαν 10 εκατομμύρια δολάρια σε Γαλλία, Μονακό και Λουξεμβούργο. Και ίσως η μεγαλύτερη ανακάλυψη που κάναμε ήταν ότι βρήκαμε 21 λογαριασμούς στην Danske Bank στην Εστονία, που ήταν υπεύθυνη για το ξέπλυμα 200 έως 230 εκατομμυρίων δολαρίων της υπόθεσης αυτής. Και μετά από αυτούς τους λογαριασμούς συνεργαστήκαμε με μια οργάνωση στην Δανία ονόματι Μπερλίνσκι που είναι εφημερίδα. Και εκεί πέρα ανακαλύψαμε ότι δεν ήταν μόνο τα 200 εκατομμύρια δολάρια που πέρασαν από την τράπεζα αυτή, αλλά πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια από τους 21 λογαριασμούς. Το άρθρο της εφημερίδας αυτής ήταν πιθανότατα το πιο δημοφιλές άρθρο στην ιστορία της δανέζικης δημοσιογραφίας. Η τράπεζα ξεκίνησε την δική της έρευνα και προέκυψε ότι όντως ε, δεν ήταν μόνο 9 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά 234 δισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν μέσα από την τράπεζα Danske και από την Ρωσία και άλλες πρώην Σοβιετικές χώρες σε ύποπτες συναλλαγές. Αυτές ήταν οι επιτυχίες που είχαμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ποιες χώρες δεν άνοιξαν έρευνες. Ήταν η Αυστρία, η Φιλανδία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, όταν ε, παραπονεθήκαμε στις αυστριακές αρχές ε, δεν ε, ξεκίνησαν έρευνα λέγοντας ότι το φορολογικό έγκλημα στην Ρωσία δεν είναι αξιόπινο, αξιόπινη πράξη στην Αυστρία. Στη Φιλανδία βρήκαμε λεφτά, προϊόντα αυτού του εγκλήματος, σε μια τρίτη φιλανδική εταιρεία, ξεπλημένο χρήμα, σε μια εταιρεία με γούνες οι οποίες γούνες επέστρεφαν στη Ρωσία. Και ζητήσαμε να επιληφθούν οι αρχές ε, της Φιλανδίας και μας είπαν ότι δεν γνώριζαν ε, αν ήταν προϊόν εγκλήματος τα λεφτά. Τον ε, Νοέμβριο του 2013 ζητήσαμε από τον Εισαγγελία στη Δανία, να σας πω, αυτό ήταν πριν έρθει στη δημοσιότητα το σκάνδαλο της τράπεζας Ντάνσκε, απέρριψαν την αίτησή μας λέγοντας ότι η επίσημη έρευνα δεν θα καταλήξει πιθανότατα σε ποινική δίωξη στην Δανία. Και έχω και δύο διαφάνειες εδώ πέρα για την άρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ερευνήσει το ζήτημα. Τέλος πάντων, επειδή ο χρόνος πιέζει, δεν θα σας πω όλες τις απαντήσεις, μόνο την τελευταία. Το 2015 ζητήσαμε από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος και μας απάντησε ότι σε αυτή τη φάση μια εγχώρια έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπο να κινηθούμε. Δεν ξέρω ποιο είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να κινηθούν από το να κάνουν μια έρευνα. Ε, έχει προκύψει όμως έκτοτε ότι το άτομο που ήταν επικεφαλής ε, της έρευνα στην αρμόδια αυτή υπηρεσία που θεώρησε ότι έπρεπε να ερευνήσει έλαβε οδηγία από του ανωτέρου του να μην το κάνει. Οπότε, από την υπόθεση Μαγνίτσκι. Καταφέραμε να βρούμε ε, τα λεφτά αυτά σε 20 χώρες. Υπάρχουν 16 έρευνες που συνεχίζονται ακόμα, 34 εκατομμύρια δολάρια που έχουν παγώσει σε 5 χώρες και 6 εκατομμύρια δολάρια που έχουν ε, επιστραφεί μέχρι στιγμής και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Συμπεράσματα, λοιπόν, από την εμπειρία μου. Το πρώτο είναι ότι οι διεφθαρμένοι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αναπτύξει ένα πολύ εκτεταμένο σύστημα ξεπλήματος ε, χρήματος με διάφορα στρώματα. Στο πρώτο είναι κάποιες ε, ρώσικες τράπεζες. Στην επόμενη φάση έχουμε Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Κυργιζία. Στην επόμενη φάση έχουμε τις τέσσερις ασθενέστερες χώρες ε, στο θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εστονία, Λιθουανία, Λετωνία και Κύπρο και τέλος έχουμε την διανομή των χρημάτων αυτών στις χώρες τελικού προορισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ Καναδά και αλλού. Ποιος ωφελήθηκε από αυτό το έγκλημα? Κοιτάξτε, προφανώς θα προκύψουν και άλλοι στο μέλλον. Έχουμε βρει 800.000 δολάρια που πήγανε στον Σεργέι Ρολντούγκιν, ο γνωστός ε, τσελίστας ε, που αποκαλύφθηκε από τα Panama Papers ότι έχει 2 δισεκατομμύρια δολάρια και θεωρείται ότι κρατάει τα λεφτά για λογαριασμό του Πούτιν. 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια απευθεία στο όνομα του Κάτσιφ, ο οποίος διώκεται στην Αμερική. Είναι ο ιό του Κάτσιφ, ο αντιπρόεδρος των ρωσικών σιδηροδρόμων και πρώην αντιπεριφερειάρχης περιφέρειας Μόσχας. 11,7 εκατομμύρια δολάρια στον Βλάνταν Στεπάνοφ, σύζυγο της Όλγα Στεπάνοβα, επικεφαλής της ΔΟΗ παριθμών 23 που έκανε την περίφημη αυτή επιστροφή και είχαμε και 266.000 ευρώ στις, στο όνομα της ατιάνας Λεξιτόβα, σύζυγο του κυρίου Λεξίτοφ, αντιδημάρχου Μόσχας. Όπως σας είπα δεν είναι πλήρης ο κατάλογος, θα αποκαλυφθούν και άλλα ονόματα στο μέλλον. Τι αγοράζουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι με αυτά τα λεφτά. Πτήσεις με ιδιωτικά αεροπλάνα, κίνητα, αυτοκίνητα, ιδιωτικά σχολεία, κοσμήματα, ενοικιάσεις ε, σκαφών ε, κτλ. Σε μια πιο εγκληματική διάσταση, τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν και για άλλους σκοπούς. Βλέπετε αυτό το περίπλοκο διάγραμμα. Πολλά από αυτά πήγαν στον Ίσα Αλζαγέντ. Ο Ίσα Αλζαγέντ είχε λογαριασμού στην ε, Κύπρο, είναι σε κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ επειδή στηρίζει το πρόγραμμα χημικών όπλων του καθεστώτος Ασάντ. Οπότε τα λεφτά τα οποία εκλάψαν από το ρωσικό κράτος χρησιμοποιήθηκαν ε, για κρυφές επιχειρήσεις του ρωσικού κράτους ε, στον πόλεμο Συρία. Θα πρέπει επίσης να επισημανώ ότι ο ίδιος μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε και για τα πλυντήρια Ρωσίας, Μολδαβίας και Αζερβαϊτζάν και τέλος μια ιδιαίτερος προβληματική περίπτωση. Αυτοί οι οποίοι ξέπλυναν τα χρήματα, στην περίπτωση Μαγνίτσκι, το έκαναν σε 10 μέρες. Εμείς έχουμε φάει 10 χρόνια σε πολλά κράτη για να καταλήξουμε σε αυτά τα συμπεράσματα και αυτό έγινε επειδή δολοφονήθηκε ο δικηγόρος μου και αποφάσισα ότι θα αφιερώσω τη ζωή μου στο να δικαιωθεί. Δεν θεωρώ ότι καμία υπηρεσία δίωξης θα μπορούσε να το κάνει ποτέ. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό ως συμπέρασμα για το ξέβλημα χρηματός στην Ένωση. Οι συστάσεις μου λοιπόν. Πρώτη σύσταση είναι επειδή ε, χρειάζεται πολύς χρόνος για να δοθούν πληροφορίες και οι περισσότερες χώρες δεν θέλουν να ξεκινήσουν τέτοιες έρευνες, θα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συλλέγει όλες τις τραπεζικές πληροφορίες ε, όχι μόνο για λόγους έρευνας αλλά και δίωξης. Πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιούνται ως στοιχεία στο δικαστήριο. Έτσι θα μπορέσουμε να φέρουμε πολλές περιπτώσεις στο δικαστήριο, κατά το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η δεύτερη σύστασή μου είναι να επεκταθεί το όριο παραγραφής. Αυτή τη στιγμή ήμουνα στην ε, Δανία, συναντήθηκα με τους εισαγγελείς εκεί πέρα και μου είπαν ότι δεν μπορούν πλέον να ασκήσουν ε, δίωξη γιατί ε, έχουν παραγραφεί αυτά μετά από πέντε χρόνια από τη διάπραξη. Δηλαδή είναι γελίο αυτό το πράγμα. Ε, γιατί αρνήθηκαν όταν πήγα το 2013 και ξεκίνησαν τώρα την έρευνα. Πρέπει λοιπόν το όριο παραγραφή να τουλάχιστον 10 χρόνια και από όταν ανακαλύπτεται το έγκλημα, όχι από όταν διαπράτεται. Και τελευταία μου σύσταση, να αντιστραφεί το βάρο του αποδείξεω. Η Ολλανδική λεγόμενη προσέγγιση στην Ολλανδία, άτομα τα οποία είναι ύποπτα για ξέπλυμα χρήματο πρέπει να αποδείξουν ότι τα χρήματά του έχουν αποκτήσει με νόμιμο τρόπο, αντί για το αντίστροφο. Και έτσι αποφεύγονται όλα αυτά τα περίπλοκα πράγματα Δηλαδή να πρέπει να πηγαίνουν ε, τα ευρωπαϊκά κράτη να ζητάνε, νομική, ε, να ζητάνε βοήθεια από το ρωσικό κράτος. Όταν απευθύνθηκε το αμερικανικό κράτος ε, για βοήθεια σε μια τέτοια υπόθεση, ο δικηγόρος ή δικηγόρος του Πρεβρεζών, η κυρία Πλέσια Τσκαγιά, έγραψε την απάντηση για λογαριασμό του ρωσικού κράτους, λέγοντας ότι δεν θα δώσουμε τις πληροφορίες και αυτό το διαπίστωσε η Αμερικανική κυβέρνηση από τα email της. Και τώρα ε, κατηγορείται για παρακόλληση της ε, δικαιοσύνης, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Και οποιοδήποτε βεβαίω απευθυνθεί στη ρωσική κυβέρνηση με τέτοιο αίτημα δεν θα λάβει καμία απάντηση. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε κύριε Μπράουντερ για την πλήρη και διεξοδική παρουσίασή σας και για τις συστάσεις σας. Ο κ. Σίρμερ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για να παρουσιάσω σύντομα την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Ασυλίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Σεργέη Μακνίτσκι και επέκεινα κατά πολέμηση της ατιμορρησίας με στοχευμένες κυρώσεις. Ε, η έκθεση υιοθετήθηκε την περασμένη Τρίτη με μεγάλη πλειοψηφία, μόνο τρεις ψήφους κατά ο εισηγητής της συνέλευσης, ο Λόρδος Ντόναλτ Άντερσον από το Ηνωμένο Βασίλειο Εργατικός, μου ζήτησε να δικαιολογήσω την απουσία του, γιατί ξόδεψε μια ολόκληρη εβδομάδα στο Στρασβούργο και τώρα έχει σοβαρή δουλειά στο κοινοβουλευτικό χαρακτήρα στο Λονδίνο. Στο νέο ψήφισμα, το, η συνέλευση υπενθύμησε το ψήφισμα 1966 του 2014 για την άρνηση της ατιμορρησίας των δολοφόνων του Σεργέη Μαγνίτσκι. Στο ψήφισμα 1966 η συνέλευση ζήτησε από τις αρμόδιες ρωσικές αρχές να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ε, πέθανε σε κράτηση ο Σεργέη Μακνίτσκι και να ε, λογοδοτήσουν οι δράστες. Όπως αναφέρεται με λεπτομέρειες στην έκθεση του Ανδρέας Γκρός από την Ελβετία και τη Σοσιαλιστική Ομάδα, ο κ. Μακνίτσκι είχε καταγγείλει μία μαζική απάτη ε, παράνομη επιστροπής φόρου εναντίον του ρωσικού ε, προπολογισμού από εγκληματίε με τη συμπεχνία διεφθαρμένων ε, αξιωματούχων. Το ψήφισμα 1966 του Ιανουαρίου του 2014 είχε σαν σκοπό στοχευμένε ε, κυρώσει εναντίον αυτών που εμπλέκονταν, με απαγορεύσει θεωρήσεων, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και προσόδων, και για να καταγγελθεί το έγκλημα και η συγκάλυψη ε, το 2014 ε, η Επιτροπή ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων θεώρησε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν έκανε πρόοδο για την εφαρμογή του ψηφίσματος και αντί να διώχθουν οι ένοχοι, οι δράστες του εγκλήματος εναντίον του κ. Μαγνίτσκι και του εγκλήματος που είχε καταγγείλει παρενόχλησαν οι ρωσικές αρχές τη μητέρα του, την Χίρα και τον πρώην περλάτη, τον κ. Μπάουντερ. Ε, η κυρία Βρασέρ, που είναι πρόεδρο τη συνέλευση, ε, διαβίβασε το ψήφισμα 1966 σε όλε τι εθνικέ αντιπροσωπείε για να δοθεί συνέχεια. Ε, την περασμένη εβδομάδα η συνέλευση σημείωσε ότι οι ρωσικέ αρχέ δεν είχαν σημειώσει πρόοδο ούτε τώρα για να διωχθούν οι ένοχοι και οι δικαιούχοι των του εγκλήματος ε, εναντίον του κυρίου Σεργέη Μαγνίτσκι και ορισμέ, όλες οι εγκληματικές υποθέσεις έκλεισαν και ορισμένοι που εμπλέκονταν, ορισμένοι υπάλληλοι κτλ. Ε, έλαβαν εφημομνία από αξιωματούχους του κράτους. Ε, και ο κύριος Μπράουντερ, ο οποίος κάνει παγκόσμια εξαρτία εναντίον της ατιμορρησίας, παρενοχλείται από τις ρωσικές αρχές. Αυτό καταδικάστηκε από τη συνέλευση σε ψήφισμα του 2017 για την καταχρηστική προσφυγή στο σύστημα του ε, Ιντερπόλ από τον κύριο Φαμπρίτσιο και την περασμένη εβδομάδα είπε ότι η Ρωσία ακόμα μια φορά αποπειράθηκε στις αρχές του μήνα να χρησιμοποιήσει με λάθος και λάθρο τρόπο τη διαδικασία Ιντερπόλ του κυρίου Μπράουντερ. Διάφορα μέρη και χώρε παρατηρητέ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπω ε, η Στονία, Λετωνία, Λιθουανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Πολιτείε, υιοθέτησαν του νόμου Μαγνίσκη που επιτρέπουν στι κυβερνήσει του να επιβάλλουν στοχευμένε κυρώσει ε, σε διώκτες και στους αποδέκτες ε, προσόδων κτλ. σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι νόμοι αυτοί ε, είναι ευπρόσδεκτοι ε, και δεν περιορίζονται σε άτομα από συγκεκριμένες χώρες ή άτομα τα οποία εμπλέκονται σε συγκεκριμένα εγκλήματα όπως ας πούμε η δολοφονία του Σαργέη Μαγνίτσκι. Την περασμένη εβδομάδα Παρακαλώ, μήπως θα μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Την περασμένη εβδομάδα η συνέλευση φέρμα καλωσόρισε την πρωτοβουλία της Ολλανδίας και άλλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσουν ένα νομικό εργαλείο που θα επιτρέπει να επιβληθούν στοχευμένες κυρώσεις σε δράστες παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναφέρει μια αναφορά στον τίτλο αυτού του εργαλείου, στον Σεργέη Μαγνίτσκι. Το όνομά του, όπως είπε η συνέλευση στο ψήφισμα, ε, είναι σύμβολο ε, και εκπροσωπεί όλους τους γενναίους ανθρώπους σε πολλές χώρες που έχασαν τη ζωή τους καταπολεμώντας τη διαφθορά, στηρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Θα ήθελα να τονίσω εκ μέρου του Λόρδου Άντερσον ότι το τελευταίο σημείο είναι τεράστια σημασία για τη συνέλευση. Το όνομα του Σεργέη Μαγνίτσκι δεν είναι απλώς ε, ένα πασίγνωστο σύμβολο στην κοινότητα που ασχολείται με τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα, αλλά είναι η μεμονωμένη περίπτωση με την καλύτερη τεκμηρίωση ε, για θέματα ατιμορρησία εναντίον σοβαρών παραβιάσεων ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, το πρώτο αίτημα της συνέλευσης ε, με το ψήφισμα του 2009, το 1685, ε, εκδόθηκε όταν ήταν ζωντανός ακόμα ο κύριος Μαγνίτσκι Και ένα άλλο ψήφισμα με έναν άλλο εισηγητή, ε, μια πράσινη ε, Γερμανίδα, ε, έφτασε στα ίδια συμπεράσματα ότι υπάρχουν σοβαρότατες παραβιάσεις με πολιτικά κίνητρα στην ποινική δικαιοσύνη. Υπάρχουν αυτή η έκθεση που έκανε ο Ανδρέας Γκρός ε, έχει πολύ λεπτομερή ανάλυση ε, εγγράφων από πολλές πηγές, από ΜΚΟ, από τη ρωσική ε, PM, υπό την UNCTAD, από δημοσιογράφους, έγγραφα, πρακτικά δικαστηρίου που δόθηκαν από τους δικηγόρους τη οικογένεια Μαγνίτσκι με τη βοήθεια του κ. Μπράουντερ. Ο κ. Γκρό έδωσε στι ρωσικέ αρχέ άπειρε ευκαιρίε να σχολιάσουν αυτά τα έγγραφα σε δύο επισκέψει στη Μόσχα όπου ε, συναντήθηκε διαμακρών με ανώτατους εκπροσώπους του Υπουργείου ε, Εσωτερικών της Ερευνητικής Επιτροπής, το αντίστοιχο ρωσικό FBI και την ε, Υπηρεσία Ομοσπονδιακών Φυλακών καθώς και τον διοικητή της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Στο ψήφισμα της περασμένης εβδομάδας η συνέλευση τόνισε τα πλεονεκτήματα των στοχευμένων, δηλαδή έξυπνων κυρώσεων αντίον ατόμων και εταιριών με τις οποίες εμπλέκονται σε αντιδιαστολή με γενικές οικονομικές ή άλλου τύπου κυρώσεις εναντίον γενικά χωρών. Ε, σε αναφορά στο προηγούμενο ψήφισμα ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, και των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους μαύρους καταλόγους κατά της τρομοκρατίας, ο εισηγητής ζήτησε από τη συνέλευση να εξασφαλίσει ότι αυτή η νομοθεσία Μαγνίτσκι θα δημιουργήσει μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία για την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων. Τέλο, η συνέλευση ζητάει πολλέ χώρε και τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν μεταξύ του για να εντοπίσουν συγκεκριμένα άτομα στόχους, να μοιραστούν πληροφορίες για άτομα τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε πίνακες ε, κυρώσεων. Νομίζω ότι έφτασα στο τέλος της, του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου. Είμαι... Τελειώνω εδώ την πανεβασή μου, αλλά μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ σημαντική αυτή τοποθέτηση. Ξεκινάει η συζήτηση λοιπόν με τους βουλευτές. Πέντε λεπτά ερωταποκρίσεις. Ένα για τον κάθε βουλευτή. Ο κύριος Νέντερμαϊερ, συνεισηγητής ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Πρέπει να πω πως είναι συναρπαστικά αυτό που μας αφηγηθήκατε, αλλά και τραγική ιστορία αφού κατέληξε ή αφού ε, έχει και τον θάνατο του κύριου, τη δολοφονία του κύριου Μακρίνσκι. βρίσκεται λοιπόν περί τα 200 εκατομμύρια ως ίχνος. Και από εκεί φτάνετε στα 200 δις που έχει νομοποιήσει η Γκτάνσκε, μικρό δείγμα διαφθοράς και εγκληματικότητας στη Ρωσία αλλά και αλλού. Και γιατί δεν ενδιαφέρεται κανείς, γιατί δεν ενδιαφέρονται οι κυβερνήσεις, γιατί πρόκειται μόνο για ιδιωτική έρευνα, γιατί όπως και να έχει όσο και αν δούμε ένα γεγονό μεμονωμένο, κάποιοι από αυτό αποκόμισαν τι δολοφονίε, δηλαδή κάποιοι αποκόμισαν χρήματα. Γιατί δεν ενδιαφέρονται οι αρχέ, λοιπόν. Επίση, δεύτερε και ε, άμεσε και ατομικέ ε, κυρώσει ε, βλέπουμε ότι φέρνουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Γιατί οι χώρε ε, διστάζουν ακόμα και σε περιπτώσει όπω το Μαγνίτσκι να αξιοποιήσουν την νομοθεσία και να επιβάλλουν κυρώσει, Ποιο είναι το πρόβλημα, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεσμεύεται στην ε, τήρηση αυτών των βασικών αξιών που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και το καθεξής. Γιατί, μα και εγώ το ίδιο διερωτώ με κάθε μέρα εδώ και δέκα χρόνια. Η απάντηση είναι πως ε, αναλόγως ο καθένας έχει διαφορετικούς λόγους να είναι επιφυλακτικό και να μην αναλαμβάνει δράση. Για να κοιτάξουμε όμως λίγο. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι ωφελούνται από τη ροή αυτή χρήματο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει πολύ ρωσικό χρήμα. Κυκλοφορεί ρωσικό χρήμα που δαπανάται και που φτάνει στα χέρια μελών του, του, του βρετανικού establishment που φροντίζουν κάποια πράγματα να μην συμβαίνουν. Βλέπουμε πληρωμές εμείς, αποδείξεις πληρωμών και σε μέλη της Βουλής των Λόρδων και αντίστοιχα άλλων. Στην ελβετική αυτή έρευνα που έχει κρατήσει εδώ και, που εδώ και 7 χρόνια από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Ελβετίας ανακαλύψαμε πως κάποιος είχε ε, σχέσεις και πληρωμές για ταξίδια στη Ρωσία από κάποιους από αυτούς. Ο αναπληρωτής Γενικός Αγγελέας της Κύπρου βρήκαμε ότι είχε μηδέουσες επαφές με κάποιους από τη Ρωσία. Αυτά είναι μόνο όσα αποκαλύψαμε εμείς. Φαντάζεστε πως είναι αυτά που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι και από την άλλη υπάρχουν και στο πιο αθώο εκείνοι που λένε ότι ε, τώρα που να τρέχω δύσκολο, που να μπλέξω με τη Ρωσία, είναι εκδικητικός ο Πούτιν, μην στρέψω τα πυρά του εναντίον μου και έτσι προτιμώ να μην κάνω τίποτα. Και μετά έχουμε και από την απλή ραθυμία. Α, κάποιος που δεν είναι και καλός στη δουλειά του, Κάποιο που μπορεί να απλώ να θέλει να χτυπάει κάρτα και να γυρνάει σπίτι του στι 5. Πάντα λέω ότι το ένα δολάριο που θα ξοδέψει για να καταπολεμήσει το κακό αξίζει όσο 100 δολάρια που θα ξοδέψει για να κάνεις το καλό, αλλά κάποιοι απλώ δεν θέλουν να καταπολεμήσει το κακό από ραφημία. Ε, το ίδιο λοιπόν και εδώ. Και σε ορισμένες χώρες βλέπουμε είτε διαφθορά, είτε ραθυμία και στον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η υπόθεση Μαγνίτσκι. Κύριο ε, Σούρμερ, και αν μου επιτρέπετε κάτι ακόμη από όλου αυτού με του οποίου είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ ω ε, εισηγητέ στην υπόθεση αυτή, ε, έχω θέσει μια ερώτηση στην οποία δεν έχω λάβει απάντηση. Ε, γιατί η Ρωσία στο ύψιστο επίπεδο των κρατικών, της κρατικής δομής και ιεραρχίας δεν αποφασίζει να διώξει τους αυτούργους του εγκλήματος, αλλά αντιθέτως ε, διώκει τα θύματα ή αυτούς που ζητούν λογοδοσία. Μια από τις εξηγήσει που ακούσαμε κατά την ε, κατάρτιση της έκθεσης Κρός ήταν και ένας από τους εισηγητές μας στην υπόθεση των Λόντρομαντ Ματ γιατί μας είπε ότι ήταν όχι νομιμοποίηση, αλλά το αντίστροφο. Ότι ο Μαγνίτσκι μπορεί να σκόνταψε απλώς στην κορφή του, παγόπουνου, του παγόβουνου της μετατροπής ποσών από τον προϋπολογισμό που υπάγονται σε έλεγχο και στη Ρωσία, όπω σε όλες τις χώρες, του Κοινοβουλίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κτλ. Μετατροπή λοιπόν αυτών ποσών σε ένα παράλληλο κονδύλιο, κρυφό προπολογισμό που αξιοποιείται για την εξαγορά ε, ε ή ισχύω σε κάποιες περιπτώσεις. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είδε το 1984 να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του, του Orwell, αλλά τον ε, σπουδαίο καινούριο κόσμο του Wells μάλλον. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ο εισηγητής μας δεν τόλμησε ποτέ γιατί δεν υπήρξαν αρκετά στοιχεία για να τεκμηριώσει μια τέτοια, ένα τέτοιο ισχυρισμό, ε, να το προβάλλει αυτό ρητά. Αλλά, και θα μας βοηθήσει εδώ και ο κύριος Διπλαμό, ο κύριος Μπρούντερ. Ε, τι άλλη λύση μπορούσε να υπάρχει. Αυτή η απάτη της φοροαποφυγής είναι πολύ συνηθισμένη. Τα 230 δις είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου. Και ο δημοσιογραφός της Νοβιακά Γκαζιέτα με τον οποίο συνεργαζόμασταν είδε ότι υπήρχαν ε, κατάλογοι σε επίπεδο εφορίας ρωσικής όλων των επιστροφών που πήγαιναν σε διάφορα γραφεία εφορίας σε ύψος ενός δισεκατομμυρίου για ένα χρόνο που έφταναν από ό,τι διαπίστωνε σε κάποιες εταιρείες που ονομάζονται μύγε, γιατί αυτές έπαιρναν τις επιστροφές φόρου και για τις διένυμαν μετά όπου δει. Η κοφή του παγόφουν δηλαδή, ήταν αυτό το οποίο ε, βρήκε κατά τύχη ο Σοπαγνίτσκι. Αυτό που δεν ήθελαν οι αρχές να εκτεθεί περαιτέρω. Όπως είπα, δεν έχουμε δει αρκετά τεκμήρια για να το αποδείξουμε, για να το στοιχειοθετήσουμε. Για άλλα πράγματα, ναι, όλα αυτά που έχουμε περιλάβει στο ψήφισμα έχουμε τεκμήρια. Γι' αυτό όχι. Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε και εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Ίσως να επανέλθουμε. Κύριο Σκόφοντ, συνεισηγητή Σοσιαλιστέ Δημοκράτε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπράουντερ και τον κύριο Σούρμερ για τι ομιλίε του. και για τον ανοιχτό τρόπο με τον οποίο μιλήσατε. Μιλήσατε δίνοντα τα ονόματα των επιχειρήσεων, των, ε, του δίκλου των λογαριασμών, των αρχών, αλλά και των ιδιωτών που κρύβονται πίσω από αυτό. Και σε αυτό χαίρομαι ιδιαίτερω ε, για τα όσα βλέπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τολμούν έχοντα γνώση να μιλήσουν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να φοβούνται για τι ε, νομικές συνέπειες κιόλα και έτσι δεν μιλούν. Σα ευχαριστώ πολύ για το θάρρο λοιπόν και το ανοιχτό πνεύμα με το οποίο μιλάτε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι για τι συστάσει σα, κύριε Μπράουντερ. Η Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία... Η Φινλανδία φαίνεται να μην θέλουν να ξεκινήσουν τέτοιε έρευνε, αλλά πέραν των όσων μα εξηγήσατε, στην περίπτωση τη Δανία, μια και είμαι και εγώ Δανό, ε, έχετε ε, έρθει σε επαφή με την Danske Bank ή την ε, αρχή δίωξη οικονομικού εγκλήματο ε, της Δανίας. Οι άλλες αντιστοιχέ αρχές ε, σα μιλήσανε και αν ναι, τι θέση ε, υιοθέτησαν για την υπόθεση αυτή. Και επίση θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με γραπτέ ερωτήσει γιατί τόσο υλικό που βλέπω και από την ε, έκθεση σα, οπωσδήποτε θα μου γεννήσει πολλά άλλα ερωτηματικά. Αλλά πάντω θα ήθελα να μου απαντήσετε σε, αυτό, ε, σε αυτά τα ερωτήματα προ το παρόν. Ο κύριο Μπράουντερ, καταρχά ξεκινώ ότι βεβαίω και πολύ ευχαριστώ να δούμε και άλλε ερωτήσει και γραπτέ, Μακάρι να μπορούμε να έχουμε μια συνεχή επικοινωνία για συνεχή ε, συμπλήρωση των στοιχείων και των απαντήσεων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία και το έγκλημα εις βάρος του και αλλά τουλάχιστον να αποτρέψουμε στο μέλλον να συμβεί κάτι αντίστοιχο και να μεριζόμαστε μόνο στα λόγια να αναλάβουμε δράση. Τώρα, σε σχέση με τις αρχές επιβολής του νόμου, αυτό που κάνουμε είναι ότι συλλέγουμε τα στοιχεία, τα περισσότερα μέσω των ε, ερευνητικών ε, εργασιών, ερευνητικών αρχών κάποιας χώρας που μετά κοινοποιείται σε άλλες ε, χώρες και έτσι ε, κοιτούμε είτε οι είτε ιδιοκτικές αρχές της, μιας, της άλλης χώρας να ενημερωθούν. και προσπαθούμε να προλάβουμε τους αυτούργους ή αυτούς που θεωρούμε αυτούργους να μην καταστρέψουν στοιχεία πάνω απ' όλα. Ωστόσο είναι δύσκολο ακόμα και για τις χώρες για τις οποίες έχουμε εξελίξει έρευνες να δείξουν ενδιαφέρον γιατί περνάνε και χρόνια ακόμα μερικές φορές και πολλές φορές και οι βουλευτές ή τα μέσα ε, είναι κάποιοι άλλοι δηλαδή οι οποίοι ε, μπαίνουν στην υπόθεση αυτή και, την, ε, και φέρνουν την αλλαγή. Με το Μπερλίνσκι ε, χρειάστηκε να περάσουν χρόνια μέχρι ότου ο τύπος της Δανίας ανακαλύψει το, την υπόθεση και προξενήσει την αντίδραση και των αρχών. Ε, συνήθως λέω και το έργο του πιο εύκολα μπαίνει στο Χάρβαρτ, στο Πανεπιστήμιο, στη νομική του Χάρβαρτ, παρά ε, εξασφαλίζει αντίδραση από τις Βρετανικές αρχές για ένα τέτοιο σκάνδαλο. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι πολύ θλιβερό αυτό, αλλά νομίζω ότι απεικονίζει την κατάσταση πιστά. Έχουμε μια πολύ ε, ψοφοδεή αντίδραση σε επίπεδο δίωξη τέτοιων εγκλημάτων στην Ευρώπη γενικά, ω κουλτούρα δηλαδή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε από την άλλη, όταν βλέπουν τέτοια προβλήματα, αμέσω ε, δράτουν την ευκαιρία, δράτουν τον της ευκαιρίας και προχωρούν. Αλλά άλλες χώρες, Γαλλία και τα λοιπά, ευρωπαϊκές, δεν θέλουν να πιάσουν ε, αυτό το καυτό κάστανο στα χέρια τους και ε, δυστυχώς δεν προχωρούν αυτές οι υποθέσεις. Έχω σοβαρές ε, αμφιβολίες για το αν η υπόθεση Ντάνσκι θα στείλει κανένα στη φυλακή. Και φυσικά αυτό, γιατί μιλούμε για πολύ χρήμα διαθέσιμο για, τους, ε, για νομοποίηση. Έτσι λοιπόν αν υπάρχει πολύ χρήμα διαθέσιμο και αν μετά η, ο κίνδυνος είναι η απόλυση, ε, το πιθανότερο είναι να, να ενισχυθούν αυτές οι τάσεις για νομοποίηση παρανομών εσόδων. Από την άλλη, αν πάει και κανείς φυλακή, μπορεί να σταματήσουν αυτές οι τάσεις. Ναι. Συγκεκριμένα ε, θέλω να... Είχατε επαφέ με Danske Bank? Όχι. Ούτε με κανέναν ε, ε, από αυτούς που καταγγέλουμε. Είναι δουλειά των αρχών να ερευνήσουν. Γκίνερ Χέκμαρκ για το ΑΕΛΚ. Έχετε δύο ευκαιρίες. Μιλήστε εσείς λοιπόν. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και για τους δύο παρουσιάσεις. Να πω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπράντερ ιδιαίτερος για τις ε, πληροφορίες μας έδωσε και για την τεράστια δουλειά που έχει κάνει εδώ και 10 χρόνια. Γιατί είναι άλλο να καταλαβαίνεις ότι κάτι τρέχει και άλλο να μάθεις το τι τρέχει ακριβώς. Και να καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα που πρέπει να μάθεις και αυτή η πτυχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Και κάνατε αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουν κάνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να προωθήσουμε αυτή την έρευνα και να δεσμευτούμε ότι θα εφαρμόσουμε έναν ευρωπαϊκό τέτοιο νόμο. Αλλά και η Επιτροπή μας ε, ακριβώς πρέπει να δεσμευτεί ότι θα ενισχύσει τα θεσμικά αυτά όργανα για να μπορέσουμε να παλέψουμε σε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο. Αυτό είναι. Το θέμα δεν είναι ε, το ξέβλημα χρήματος που ούτως ή άλλως ε, βεβαίως ε, είναι επιλήψιμο, αλλά υπάρχει μια διάσταση η οποία απειλεί την Ευρώπη και τις δημοκρατίες μας. Ελπίζω λοιπόν να συμφωνούμε όλοι στο τι πρέπει να κάνουμε. Να θέσω και ένα ερώτημα. Νομίζω το είπατε και εσένα. Αλλά και πάλι. Είναι σαφές ότι κανείς στην Ρωσία δεν έχει ερευνηθεί και διωχθεί για τις ε, εγκληματικέ αυτές πράξεις. Μία ερώτηση είναι αυτή. Μία δεύτερη που αφορά και τους δύο σας αλλά ίσως ιδιαίτερα τον κύριο Μπράντερ θα θέλατε να επεκταθείτε στις απειλές ασφαλείας που προκύπτουν από αυτά τα τεράστια ποσά. Αναφερθήκατε στο θέμα της Συρίας. Πρέπει όμως να έχουμε μια ευρύτερη αντίληψη του ποιο είναι το θέμα. Καλό θα ήταν να μας πείτε πώς ακριβώς βλέπετε τις ε, αδυναμίες τα ανέφερε και ο Δανός ε, συνάδελφος. Γιατί δεν είναι κάτι αξιόπινο. Επειδή το καταλαβαίνουν οι αρχές ή είναι έλλειψη νομοθεσίας ή δεν υπάρχει αντίδραση. Επίσης θα ήθελα να μας ε, πείτε και το είπατε και στην ε, παρουσίασή σας ε, ποια είναι τα δύναμα σημεία, η δύναμη κρίκη στην Ευρώπη. Αναφέρατε κάποιες χώρες, την Κύπρο, θα θέλατε να εξηγήσετε γιατί ε, είναι αυτές οι χώρες ε, αδυναμικρικοί. Όλοι έχουμε κάποια ιδέα, αλλά καλό θα ήταν ε, να μας τα πείτε. Και μετά. Η άποψή σας για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε όσον αφορά την υλοποίηση του νόμου και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη, στην υπατή εκπρόσωπο, σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δράσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσένα. Σύντομα, υπήρχαν κάποιες έρευνες κατά κάποιων χαμηλόβαθμων ε, αξιωματούχων στι ε, φυλακές ε, για αμέλεια στην περίπτωση μαγνητική αλλά δεν κατέληξαν πουθενά. Και περιγράφονται μάλιστα στην έκθεση ότι κανείς ε, δεν τιμωρήθηκε. Επίσης, η κοινοβουλευτική διάσκεψη κατέληξε πρόσφατα σε μια έκθεση για το ξέπλυμα χρήματος ε, και τα σχετικά αυτά προϊόντα του εγκλήματος και μάλιστα ζητάμε από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν το Ολλανδικό μοντέλο, το Ιρλανδικό όπως λέγεται, την αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως για να υπάρχει δίμευση χωρίς ε, καταδίκη. το μοναδικό εργαλείο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί έχω σε είμαι σε επαφή με εισαγγελίε που είναι κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή και, και από τη χώρα μου τη Γερμανία που πραγματικά απογοητεύονται από το πόσα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να έχουν για να δημεύσουν το οτιδήποτε. Γιατί υπάρχει μια λάθος αντίληψη της προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας που βασίζεται και στην ε, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό όμως δεν προστατεύει τα προϊόντα εγκλήματος. Οπότε έχουμε την δυνατότητα εδώ πέρα να έχουμε πάρα πολύ ισχυρά εργαλεία για την ιδιοκτησία εγκληματιών και διεφθαρμένων. Αυτό το οποίο θέλουν, ε, τα λεφτά δηλαδή. Αυτά θα δώσουν στους εγγελεί τα εργαλεία που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά του. Αλλιώ θα το παρατήσουν. Θα ξεκινήσω με το ερώτημά σας ε, για το τι κίνδυνο αντιπροσωπεύει αυτό το ξέπλυμα χρήματος. Πολλοί θεωρούν ότι είναι κάτι το ανώδυνο, ένα έγκλημα χωρίς θύμα. Δεν ισχύει αυτό. Το θύμα εδώ προφανώς ήταν ο Σεργέη Μαγνίτσκι, αλλά υπάρχει κάποιο άλλο θύμα. Η διαφθορά της Ευρώπης. Ανέφερα τον Ελβετό αστυνομικό, τον ε, αναπληρωτή Γενικό της Κύπρου, μέλη της Βουλής των Λόρδων, που έλαβαν χρήματα από αυτούς τους εγκληματίες. Και έχουν ε, διαφθαρεί άρα και για κάθε έναν που βρήκαμε εμείς θα υπάρχουν άλλοι 10 που δεν βρήκαμε. Ανέφερα τι πληρωμέ στον Αλζαγέντ, ο οποίο ε, είναι γνωστό ότι είναι υπεύθυνο για την ε, στήριξη του προγράμματος χημικών όπλων του Συριακού Καστότος. Για το από βρήκε τα συγκεκριμένα λεφτά δεν το ξέρω ε, και το τι θα τα κάνει, αλλά φαντάζομαι δεν το δώσανε για καλό. Όπως ανακάλυψε ο Ρόμπερτ Μίλλερ, ε, τα βρώμικα χρήματα από την ε, Ρωσία πήγαν στο Facebook και στο Twitter για να χειραγωγήσουν τις αμερικανικές εκλογές. Μιλάμε μια πολύ βρώμικη υπόθεση που επεκτείνει τους στόχους ε, του Πούτιν που θέλει να προκαλέσει διχόνοια και χάος στην Δύση και το κάνει με αυτά τα λεφτά. Και αν δεν τα σταματήσουμε θα συνεχίσει. Όσον αφορά τώρα τους αδύναμους κρίκους. Ε, χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος, ε, θα χρειαζόταν ώρες. Και να αφαιρθώ σε κάποια έτσι γνωστά. Η Κύπρος είναι πολύ αδύναμος κρίκος. Χρειάστηκαν πάνω από δύο χρόνια για να απαντήσει στο αίτημα του Γάλλου ανακριτή για τραπεζικά έγγραφα. την στιγμή που δεν συνεργαζόταν μαζί του, συνεργαζόταν με την ρωσική κυβέρνηση και επέτρεπε σε Ρώσους αστυνομικούς να έρθουν στα γραφεία της εταιρείας μου στην Κύπρο. Δεν συνεργαζόταν δηλαδή με τις ευρωπαϊκές διοκτικές αρχές, αλλά με τις ρωσικές για να με διώξουν εμένα. Γιατί είναι εξωφρενικό και δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να τιμωρηθεί επειδή δεν συνεργάζεται ε, με τις ε, νόμιμες διοκτικές αρχές. Ε, γιατί το κάνει τώρα. Μάλλον για τον ίδιο λόγο που είδαμε ότι είχε επηρεαστεί ο ανοπλωτής Γενικός Αγγελέας. Πολλά λεφτά πάνε στην Κύπρο και πολλοί κόσμος ζει από αυτή την υπόθεση και έχει τελείως αντικρώμενα συμφέροντα. Και μιλάμε επίσης ε, για τον νόμο Μαγνίτσκι. Πέρασα 9,5 χρόνια. Ε, τώρα, 6 χώρες έχουν τέτοια νομοθεσία. Ηνωμένε Πολιτείες, Καναδάς, ε, Ηνωμένο Βασίλειο και οι τρεις Βαλτικές. Ε, από την αρχή έχω προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018 πέρασε ένα ομόφωνο ψήφισμα εδώ πέρα για να πέρασει ένα τέτοιο νόμος και η επικεφαλής ε, της Υπηρεσίας εξωτερική Δράσης, η κυρία Μογκερίνη, το απέρριψε. Απέρριψε αυτό το αίτημα και τα επόμενα αίτηματα. Και μας είπαν ότι αν θέλετε να περάσετε τέτοια νομοθεσία πρέπει να πάτε στο επίπεδο των κρατών μελών. Πήγαμε λοιπόν στα κράτη-μέλη και μας είπαν ναι, είναι καλή ιδέα, αλλά πρέπει να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ένας φιλικός βουλευτής στην Ολλανδία μας είπε, ωραία, να το κάνουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να περάσουμε ένα ψήφισμα εμείς στο δικό μας κοινοβούλιο, το Ολλανδικό. Και το ΒΒΔ στην κυβέρνηση είπε, α, όχι τώρα, που τι να κάνουμε. Και επειδή ήταν κυβέρνηση μειοψηφία, ε, το ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι και το πέρασαν. Και ζήτησαν από την Ολλανδική κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Στέφαν Μπλοκ, ο Υπουργό Εξωτερικών, μετά υπέβαλε μια πρόταση στο ευρωπαϊκό επίπεδο και έσβησε το όνομα Μαγνίτσκι από την πρόταση και είπε σε διάφορες Ολλανδούς βουλευτέ εδώ πέρα μην αναφέρουν το όνομα του Μαγνίτσκι. Γιατί? Για να κατευνάσει τη Ρωσία. Ε, είναι ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα. Και ένα από του στόχου μου σήμερα εδώ πέρα, πέρα από την κατάθεσή μου εδώ, είναι ακριβώς να βρω στήριξη από όλε πολιτικές ομάδες για ένα ψήφισμα που θα ζητάει από την Υπηρεσία εξωτερική δράση να ξαναμπεί το όνομα του Μαγνότσκι όπως έχει μπει και σε όλες τις άλλε χώρες. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ε, έχει επικυρώσει αυτό το αίτημα λόγω της συμβολικής ε, φύσης του ονόματος του Σεργέη Μαγνίτσκι, όπως είπα και στην παρουσίασή μου κύριος Χόκμαρτ, ε, εκτός μικροφώνου. Η Άννα από τους σοσιαλιστές. Γιατί κατά την απόψή σας υπάρχει αυτή η αντίσταση για να έχουμε στην Ευρώπη ένα νόμο αντίστοιχο με το Μαγνίτσκι. Ε, κάτι που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα το 2013, ε, με το όνομα Μαγνίτσκι τότε. Τότε το είχαμε συνδέσει με τον αγώνα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ε, κύρωση εκείνων που είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις τους. Αλλά πολύ περισσότερο τώρα για να καλύψουμε και αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι η καταπολέμηση του ξεπλήματο του χρήματο. Μακάρι ο Γκούνερ Χόκμαρκ να ήταν ο εκπρόσωπο του ΕΛΚ. Από αυτά που είπε σήμερα, για αυτή την υπόθεση μου άρεσε. Πολλές από τις προτάσεις ε, που έκανε ε, τις μπλόκαρε το ΕΛΚΑ και οι διάφορες κυβερνήσεις, του, οι δεξιές. Κυρίως την πρόταση για ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος σε κεντρικό επίπεδο ε, σε Ευρωπαϊκή Ένωση μία ευρωπαϊκή υπηρεσία, ας πούμε, καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος ε, που θα συνεργάζεται με την Eurojust. Με αναφερθήκατε σε αυτή τη δικηγόρο, η οποία παράλληλα ε, με, την, με τις επαφές με τον Τραμπ συνέτασε και την απάντηση που έδωσαν στους Αμερικανούς εισαγγελείς. Μιλάμε για εξαγορά ε, ανθρώπων. Αυτό, κάτι αντίστοιχο, μπορεί να συμβαίνει και στις χώρες, στις δικές μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά. Μπορείτε να το σχολιάσετε. Επίσης, είπατε ότι το ίδιο πλυντήριο που χρησιμοποιήθηκε για το ρωσικό χρήμα, χρησιμοποιήθηκε και για μολδαβικό και αζερικο χρήμα. Το γεγονός ότι, όπως υπόθηκε, τα κράτη-μέλη δεν ε, συνειδητοποιούν ότι η διαφθορά είναι μορφή υβριδικού πολέμου, ίσως αν σας ακούσουν ε, να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία για, τα, για, τους Ρώσους. Ε, μπορεί να ασχοληθούν περισσότερο με τους Ρώσους και όχι με τους Μολδαβούς ή ε, Αζέριους. Τα πλυντήρια αυτά ξεπλήματος δεν γνωρίζουν γεωγραφικές διαφορές ανάμεσα στους εγκληματίες. Όλοι αυτοί συνεργάζονται. Ξεπλένουν χρήμα μαζί, παίζουν μαζί. Όλοι χρησιμοποιούν τους ίδιους δικηγόρους, τα ίδια καταπιστεύματα, τους ίδιους τραπεζίτες, ίδιες τράπεζες. Το σύστημα είναι πάρα πολύ εξελιγμένο. Όσο μπαίνει κανείς σε λεπτομέρειες για τέτοιο ξέπλυμα, πρέπει να έχεις τέτοια προσοχή, τέτοιες ε, γνώσεις, που βλέπεις ότι όταν δημιουργηθεί αυτό σωλήνα, σε αυτά τα κανάλια, ας πούμε, όλοι τα χρησιμοποιούν. Γιατί αυτό είναι πολύ άσχημο, γιατί χρησιμο... Ε, περνάνε πολλά λεφτά από εκεί, αλλά είναι και καλό γιατί άπαξε το ανακαλύψαμε, το εκθέτουμε. Και το εκθέτουμε πώς. Χρησιμοποιώντας ε, κάποιες ε, κάποια νήματα, α πούμε, παραδείγματος χάρη την υπόθεση Μαγνίτσκι, την έρευνα, ας πούμε, ε, στο Αζερβαϊτζάν και μπορούμε να διαλύσουμε αυτό το κανάλι. Βεβαίω μπορούν να χτίσουν νέα κανάλια οι εγκληματίες αυτοί, αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να το φτιάξουν εάν κάνουμε κάτι από αυτά για τα οποία μιλάμε σήμερα. Αν κάποιε αυτέ τι υποθέσει, α πούμε, φτάσουν στα δικαστήρια. Κάποιοι από αυτού του νόμου αρχίσουν να εφαρμόζονται. Ένα από τα βασικά θέματα εδώ είναι η έλλειψη εφαρμογής. Ε, σίγουρα θα πρέπει να αλλάξουν και οι νόμοι, το συζητήσαμε. Αλλά ακόμα και να αλλάξουν όλοι οι νόμοι, εάν δεν εφαρμοστούν οι νόμοι, εάν δεν αρχίσουν οι διώξει, εάν δεν αρχίσουν οι παραπομπές στα δικαστήρια και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, δεν θα πρέπει να αισθανθεί κανένα φόβο, α πούμε, από αυτήν την ιστορία. Οι άνθρωποι δηλαδή που θα πρέπει να φοβούνται. οι διοκτικέ αρχές των ε, κρατών μελών θα πρέπει να ασχοληθούν. Ε, είδα το Ηνωμένο Βασίλειο και είδα πόσο σοκαριστική είναι η κατάσταση του Ηνωμένου Βασίλειου. Δεν θα πω ότι Έχουμε πάει πέντε φορέ, ας πούμε, στι διοκτικέ αρχέ στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, για τα θέματα τη υπόθεση αυτή και δεν κάναν τίποτα, α πούμε. Στο Κοινοβούλιο επίση. συχνά ε, οι πολιτικοί λένε θα κάνουμε κάτι, αλλά οι διοκτικές αρχές που εκφεύγουν του, του πολιτικού ελέγχου και δεν είναι κάτω από πολιτική πίεση, ας πούμε, αποφασίζουν να μην κάνουν τίποτα. Είναι σαν να οδηγεί, πούμε, ε, ένα αυτοκίνητο και δεν έχεις κανένα έλεγχο ας στο τιμόνι. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε και να, να κρατηθούμε από οτιδήποτε. Την τροπή, ε, τις σχέσεις, ε, τις διαπλοκές κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, διστάζω να ε, συμφωνήσω με την ιδέα ότι πρέπει η τήρηση και επιβολή του νόμου να τεθούν υπό τον έλεγχο της ε, εκτελεστικής εξουσίας και η ερμηνεία τους βέβαια. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να μην χαθεί η διάκριση των εξουσιών αλλά η τήρηση οπωσδήποτε του νόμου πρέπει να εξασφαλίζεται. και μάλιστα κατά τρόπο διαφανή ώστε να μην προσκρούμε σε τείχο όπως συμβαίνει πολλές φορές τώρα για την έκθεση για τη διευκόλυνση δημεύσεως παρανομών ασόδων. Πρέπει αυτό να γίνει στην Ευρώπη. Το έχουμε ζητήσει και έχω πει επανελειμμένως ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπήρχε ένα μητρό κεντρικό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. γιατί τα μεμονωμένα μητρώα των κρατών είναι ισχνά, πολύ ισχνά. Και στη Μάλτα και στη Γερμανία είδαμε ότι οι αρμόδιες αρχές, να, το σκάνδαλο στη Γερμανία με τους τελωνιακούς. Εκεί πρέπει να ενισχυθεί η διάσταση της επιβόλης του νόμου. Κυρία Γκόμες, έχει προταθεί, ξέρετε, από την έκθεση τάξη που υιοθέτει στο Κοινοβούλιο ένα ευρωπαϊκό FIU και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση των, της νομοποίησης εσόδων, αλλά κάποιες, κάποιες κυβερνήσεις απέρριψαν την ιδέα αυτή από το Συμβούλιο. Ο κύριος Γιζεκ, ναι, αλλά θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και ελπίζουμε ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. κυρία Σκοτ Κέιτο, πράσινη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε κατάθλιψη αισθανόμαστε όταν ακούμε όσα έχετε να πείτε καταγράφοντας τις αδυναμίες και την ε, αδιαφορία ή την απουσία βούλησης ε, και για τη δική μου τη χώρα συγκεκριμένα που επιτρέπει στην ε, Ρωσία να κάνει αυτή, αυτά που κάνει. Έχω ένα website όπου καταγγέλλω τους bad boys του Brexit, τα κακά παιδιά του Brexit και βεβαίως ε, τις δραστηριότητες για χειραγώγηση του πολύ κακού, όπως πιστεύω εγώ, δημοψηφίσματος. Εγώ είμαι από το Κλώστερ που είχαμε και δολοφονία έως και 14 θανάτους ύποπτους που δεν έχει διερευνήσει επαρκώ η αστυνομία. Υπόπτους ε, και πιθανόν να έχουν υποκινηθεί από τη Ρωσία. Άρα τα θέματα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο σε οικονομικούς όρου, αλλά και σε όρου εθνική ασφάλειας. για την υπόθεση τη εισαγωγή νομοθεσία τύπου Μαγνίτσκι. Το πρόβλημα που έχω εκεί εγώ είναι ότι αυτή η νομοθεσία, αυτό ο νόμο απαιτεί απόδειξη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Ολλανδοί έχουν περάσει αντίστροφα και έχουν ανατρέψει την ε, το βάρος της απόδειξης. Αλλά όταν έχουμε πολύ περίπλοκα συστήματα νομοποίηση παρανομών εσόδων. Είδαμε και με τις δολοφονίες των δύο ε, Ρώσων στην ε, Βρετανία. Γιατί αντί να αφήνουμε να μπαίνουν τα χρήματα αυτά να μην ζητούμε από οποιονδήποτε έχει να φέρει χρήματα να αποδεικνύει ότι είναι της νομοταγή και ότι καλά κάνει και φέρνει τα χρήματα και έχει και το Απάντηση Μπράουντερ, ευχαριστώ. Ε, θεωρητικά πρέπει, οφείλει κάθε τράπεζα να ζητεί θεμητή αιτία συναλλαγή. Αυτό απαιτούν όλοι οι κανονισμοί για την καταπολέμηση των, παρα... της νομοποίησης παρανομών εσόδων ε, που είναι να γνωρίζει δηλαδή η τράπεζα ποιος είναι ο πελάτης της. Λοιπόν, να σας πω ένα πολύ απλό. Ε, πρέπει κανονικά πάντα να γίνεται ο έλεγχος των εσόδων. Έτσι, εγώ έχω δημοσιεύσει ένα βιβλίο που λέγεται Red Book, η Simon και Schuster ε, είναι ο εκδοτικός μου οίκος, μου πληρώνουν 12.000 δολάρια για τα πνευματικά δικαιώματα και η HSBC η τραπεζά μου όταν φτάνουν τα λεφτά αυτά στο λογαριασμό μου, μου παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει να σου πω αυτό ο Σιμών Σουστέρ, τι ποιο είναι που σου στέλνει λεφτά. Και λέω, Όχι, είναι ένα πολύ γνωστό εκδότη και μου πληρώνει τα πνευματικά μου δικαιώματα κτλ. Με ενοχλεί λοιπόν να πρέπει η τράπεζα να ελέγχει τα 12.000 που παίρνω εγώ ω αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα και να αφήνει να περνούν από τεράστια παράθυρα που υπάρχουν στην νομοθεσία ποσά δισεκατομμυρίων. Και βέβαια να μην, να μην προβλέπονται καν κυρώσει αυτή τη στιγμή. Για το βάρος απόδειξης και τις κυρώσεις. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ο νόμος Μαγνητσκή στην παγκόσμια εκδοχή του τιμωρεί και την ομοποίηση και τους κλεπτοκράτες. Η πρόταση του Ολλανδού Υπουργού για Ευρωπαϊκό νόμο Μαγνίτσκι, που δεν θα έχει το όνομα Μαγνίτσκι όμως, αναφέρεται μόνο σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει μόνο μία προσθήκη, ότι δηλαδή ευθυγραμμίζεται στον Αμερικανικό ή Καναδικό ή άλλους αντίστοιχου νόμους για να καλύψει και την κλεπτοκρατία. Αλλά είναι βαρύ το βάρο απόδειξη. Φυσικά και πρέπει να είναι, δεν πρέπει δηλαδή με το παραμικρό κάποιο να μπαίνει στη λίστα αυτή ε, και πρέπει να διώκεται και η παραβίαση των δικαιωμάτων και η νομοποίηση. Για το βάρο απόδειξη νομίζω ότι έφερα εγώ τα επιχειρήματά μου, όπω και το Συμβούλιο τη Ευρώπη, και νομίζω ότι είναι απλό. Μια απλή λύση δηλαδή, ότι όταν υπάρχουν κάποιες ε, ύποπτε συναλλαγέ, πρέπει να αποδεικνύεται ότι δεν είναι ύποπτε. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ε, εισαγάγει νόμο που λέγεται Unexplained Wealth Orders, δηλαδή ε, εμβάσματα χωρίς πόθεν έσχε. Ναι, ένα λεπτό που σας διακόπτω, συγγνώμη. Δηλαδή κάθε μεγάλη συναλλαγή θα πρέπει να γίνεται από τη Ρωσία, θα πρέπει να γίνεται, να θεωρείται ύποπτη. Ε, δεν θα διαφωνήσω απαραίτητα μαζί σας. Ίσως ο κύριος Σούρμερ. Ναι, όχι, εγώ θα διαφωνήσω. Δεν μπορεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που έρχεται από τη Ρωσία να είναι ε, παράνομη. Έχουμε εξαγωγές φυσικού αερίου, πετρελαίου, πρέπει να πληρωθούν ε, ε, οι τιμές αυτές, ε, θεμητό εμπόριο, ούτε και κάθε πράξη των αρχών της Ρωσίας ή των δικαστηρίων της είναι πράξη που υποκρύπτει διαφθορά. Αλλά υπάρχει μια ηγεσία, μια ελίτ, έναντι της οποίας πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, γιατί έχουμε έστω ανεκδοτολογικά πολλά περιστατικά, και τα έχω δει εγώ στα δρομία μου, χειραγώγησης και των αρχών τήρησης του νόμου και των δικαστικών διαδικασιών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οτιδήποτε δούμε να προέρχεται από τη Ρωσία αυτόματα θεωρείται παράτυπο ή παράνομο. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει κάθε συναλλαγή που προέρχεται από τη Ρωσία να διερευνάται ως ε, ε, ύποπτη. Αντίστροφα όμως θα πω ότι κάθε συναλλαγή που ξεπερνά ένα όριο ελάχιστο Να, να σας πω ο γιος μου που πήγε να ζήσει στο εξωτερικό χρειάστηκε να φτιάξει το σπίτι του για, και για να το αγοράσει εγώ τον ε, βοήθησα όταν έστειλα ε, εγώ τα χρήματα χρειάστηκε στο έμβασμά μου να βάλω και μια υποσημείωση που έλεγε ότι να δουλεύω τόσα χρόνια, έχω μαζέψει τα λεφτά αυτά ως αποταμίευση και τα δίνω ως δάνειο στο γιο μου για να στήσει το σπιτικό του. Ωραία λοιπόν, γιατί να μην ισχύει αυτό κι αλλού, χωρίς διακρίσεις ε, προελεύσεως, χώρας κτλ κάθε συναλλαγή που θα ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να επαληθεύεται ως προς την έστω πρίμα φάκη νομιμότητά της. Και το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν ζητεί την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης για την επιβολή των κυρώσεων, αλλά για το πάγωμα των ε, παράνομων ή των ύποπτων εσόδων. Αυτό παρακαλώ για να είναι σαφές. Για τις κυρώσεις δεν μπορεί να έχουμε τις, ε, δεν μπορούμε να έχουμε βάρος απόδειξης διαφορετικό και να ξεπερνούμε την ε, επαρκή τεκμηρίωση ή υποψία για την επιβολή τους και ταυτόχρονα πρέπει ο υποπτός να έχει την ευκαιρία να απαντήσει, να ανταποκριθεί και να δώσει εξηγήσεις. Αυτό άλλωστε το έχουμε και στην έκθεση του Λόρδου Άντερσον. Για να μην ε, βγει καμία ε, παρεξήγηση από τα όσα είπα. Φυσικά το κράτος δικαίου ισχύει και πρέπει να ισχύει και για εκείνους που καταπολεμούν όσους παραβιάζουν το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ, Νικόλα Μπή. Ευχαριστώ. Στι 27 Απριλίου του 2016 και κατόπιν προσκλήσεως φιλανδή βουλευτού, ο Αντρέι Νεκράσοφ, σκηνοθέτη και γνωστό για την στράτευσή του για την καταπολέμηση αυτού που ονομάζει σύστημα Πούτιν, ερχόταν να παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώ την ταινία την αφιερωμένη στην υπόθεση Μαγνίτσκι. Να μια πρώτη κύρωση λοιπόν από τα ευρωπαϊκά κράτη για τη Ρωσία και θα έπρεπε μετά να βγει και στι 3 Μαου στο Άρτε. Λίγο μετά, τελευταία στιγμή όμω. Ε, βγήκαν από το πρόγραμμα οι δύο αυτές εκδηλώσει, ακυρώθηκαν, ε, λογοκρίθηκαν και στο κοινοβούλιο, δηλαδή και η προβολή του Άρτε, ενώ το, ε, η ταινία αυτή που είχε συγχρηματοδοτήσει το Άρτε είχε περάσει όλα τα κριτήρια επαλήθευση της αξιοπιστίας της. Γιατί λοιπόν αυτή η λογοκρισία σε μια, λογοκρισία γεωγραφική περιοχή όπου υποτίθεται πως ε, επικρατεί η απόλυτη ελευθερία και δημοκρατία ο Νεκρασόφ καταρχάς προσέφερε τις εξηγήσει της αντίστοιχης με τον κύριο Μπρόντερ, Μπράουντερ. Ωστόσο μετά έκανε και τη δική του έρευνα ε, για να δει τι είχε συμβεί για όλους εκείνους που δεν είχαν ε, λάβει το λόγο. Έτσι λοιπόν η αίσθηση του κυρίου Μπρόντερ ανακαλύψει ο κύριος Νεκρασόφ ότι είχε κάποια στοιχεία παρουσιάσει τα οποία ήταν έως και ψευδή όπως μια φωτογραφία ενός νέου που είχε υποτίθεται κρατηθεί σε νοσοκομιακή ε, πτέρυγα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ναι, ένας νεαρός είχε ξυλοκοπηθεί από τους Αμερικανούς, αλλά ήταν στις Ηνωμένε Πολιτείε και δει το 1961, κύριε Μπρόντερ, η φωτογραφία που δείξατε. Ε, άρα λοιπόν εδώ μιλούμε για δυσφήμιση και εφόσον σας το αναφέρω εδώ μπορείτε να κάνετε και στον κύριο Νέκρασοφ τη σχετική μήνυση για τσικοφαντική δυσφήμιση. Αλλά ο κύριος Νέκρασοφ ταυτόχρονα 13 Νοεμβρίου έκανε και μάλιστα στο τοπό του υπάρχει και η σχετική ανάρτηση και όλα τα στοιχεία, δεν χρειάζεται να πιστεύουμε μόνο σε αυτά που λέει αν δεν έχει τεκμήρια. Ε, και όπω είπα, μπορείτε να του κάνετε σκοφαντική, για σκοφαντική δυσφήμιση. Έχει δώσει λοιπόν όλα τα στοιχεία για τι δυσκολίε που αντιμετώπισε στην ετοιμασία αυτή τη ταινία. Κύριε Μπράουντερ, σε όλο τον κόσμο εσεί ε, δηλώνετε πω είστε ο υπαριθμόν ένα εχθρό του Βλαντιμίρ Πούτιν και αυτό εντό εισαγωγικών γιατί είναι δικά σα λόγια. Θα ήταν, θα ήταν ε, ε, περιγέλαστο αν δεν ήταν τόσο σοβαρά και τραγικά τα πράγματα. Ρωτώ λοιπόν συγκεκριμένα δεν είναι τώρα η η στιγμή να έρθουμε σε μια καταντιμολία αντιπαράθεση μεταξύ ημών κύριε Μπρόντερ και του κυρίου Ντέμπρασοφ, ο οποίο τελευταία ανάλυση εκλήθη να μαρτυρήσει στο ε, Κογκρέσο των ΗΠΑ και μάλιστα κανεί δεν του μίλησε για σκοφαντική δυσφήμιση ούτε του έκανε μήνυση. Κύριε Μπρόντερ, για να απαντήσετε. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ε, φανταζόμουν ότι από το FSB θα υπήρχε κάτι και πολύ ευχαρίστως να δώσω απαντήσεις. Αν είναι εδώ το FSB, πολύ ευχαρίστως να σας δώσω την απάντησή σας λοιπόν. Ο Νέκρασοφ είναι ένας ύποπτος σκηνοθέτης, κάνει ψηλοδουλίτσες για τον Εμπερεζόφσκι κατά του Πούτιν, ταινίε και όταν έκανε παλιά και όταν, όταν πέθανε ο Εμπεριζόφσκι, του τέλειωσε το χρήμα και έτσι χρειάστηκε νέο χορηγό ο οποίος ήταν το FSB πρώην KGB της Ρωσίας από ό,τι ξέρω εγώ Έτσι λοιπόν ο Νεκρασόφ ετοίμασε μια ταινία προπαγάνδας με το FSB, με ό,τι του είχαν υποδείξει, να περιλάβει και προσπάθησε σε κάποιες περιπτώσεις να προβάλλει την ταινία του. Εμείς όμως ε, φέραμε αντιρρήσεις, γιατί αυτή η ταινία είναι πλήρης ψευδών και παραπληροφόρηση. Μερικέ φορέ να έγινε και δεκτή η επιφύλαξή μα, όπω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά σε περιπτώσει έγινε προβολή τη ταινία, όπω στη Ουάσιγκτον, όπου όσοι την είδαν αντελήφθησαν ότι ήταν μόνο ρωσική προπαγάνδα αυτή η ταινία. Δεν θεωρώ ότι είναι ο Νεκράσοφ δικηγόρος, τίποτα άλλο παρά όργανο της προπαγάνδας και δεν πρόκειται να κατεβώ το επίπεδο του για να έρθω σε συζήτηση μαζί τους, καμία περίπτωση. Κύριο Σούρμερ, ναι, θα προσθέσω ότι αυτή η ταινία το 2016, του 2016 εξετάστηκε στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να κριθεί ως ένα κατάφορο παράδειγμα παραπληροφόρησης. Ο πρώτος αντιπρόεδρος Φαμπρίτσιο ήταν και στο ε, διοικητικό συμβούλιο στη Γερμανία για το θέμα αυτό και με τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας και τα τεκμήρια μπορέσαμε να του εξηγήσουμε ότι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά παραπληροφόρηση αυτή η ταινία. Ξέρω πολύ καλά λοιπόν και με αρκετές λεπτομέρειες ότι κάποιες, ε, πώς ε, παρήχθησαν ορισμένες από τις σκηνές του ταινία ο Νέκρασοφ. Ξέρω ότι επετέθη λίγο πολύ με ένα μικρόφωνο και μια κάμερα στον Ανδρέας Γκρό, τον πρώην εισηγητή μου, κραδένοντα ένα κομμάτι χαρτί στα ρωσικά, ε, ισχυριζόμενος πράγματα που δεν ισχύουν χωρί καν να επικαλείται κάποιον συγκεκριμένο. Ο κύριο Μαγνίτσκι ποτέ δεν κατηγόρησε κανέναν, ε, ούτε τον αστυνομικό που τον είχε προφυλακίσει ούτε κανέναν άλλον συγκεκριμένα. Ήταν λάθος, ψέματα όλα αυτά. Κατάφορα ψέματα. Μετά αυτό το χαρτί που είχε δοθεί στον κύριο Γκρός το εξετάσαμε στη μετάφρασή του από τα ρωσικά αλλά και στα ρωσικά απευθεία και είδαμε ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια να παγιδευτεί ο κύριο Γκρός όπως και η κυρία Μαρή Λουίς Μπέκ στο Βερολίνο, στο γραφείο της, όταν κατηγορήθηκε από τον κύριο Νέκρασοφ ότι, είναι, ότι έχει ένα βοηθό που στην πραγματικότητα ε, είναι πράκτορα στη CIA και σε μένα είχε έρθει στο Στρασβούργο, στο γραφείο μου, προσπάθησε να μπει μέσα αλλά δεν τον άφησα. Έχω εξοργιστεί με αυτή την ιστορία και θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για αυτή την ε, πίθανη προπαγάνδα. Μην σας κουράζω με τις λεπτομέρειες, αλλά κύριε Μπέ, πολύ ευχαριστώ να σας δώσω τις πληροφορίες. Γιατί μια και είχε ήδη ε, συνταξιοτηθεί ο εισηγητής, ο πρόεδρος τότε ήταν απολύτως αποφασισμένος να μην μείνει παραμικρή σκιά προ την ακαιρεότητα της επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επιτροπή μας δεν έχει αρμοδιότητα να ασχολείται με ταινίε. Ε, είτε από πλευρά περιεχομένου είτε από πλευρά καλλιτεχνικής αξίας. Έχουμε ένα αίτημα από τον κύριο στρεβίτσης για να μιλήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, το θέμα δεν αφορά την καλλιτεχνική αξία ταινιών, αλλά στη συγκεκριμένη στιγμή εδώ μέσα δεν θα πρέπει να ακούγονται ψευδείς ειδήσει και ψέματα. Ίσως δεν θυμούνται πολύ εδώ μέσα την ημέρα που θα έπρεπε να δούμε την ταινία του κυρίου Νεκάσοφ και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τον ακολουθούσε η κυρία Βυσεβίτσικα για η οποία είχε συναντήσει τον Ντόναλτ Τραμπ πριν από τις εκλογές και ήταν ειδική εκπρόσωπος ε, του Κρεμλίνου στην ομάδα του Τραμπ. Ε, είναι δύσκολο βεβαίω να είναι κανεί ανεξάρτητο όταν το κόμμα το χρηματοδοτούν οι ρωσικέ τράπεζε και γύρονται διάφορα ερωτήματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δύο Ρώσοι κατάσκοποι έκαναν την δολοφονία στο Σόλσβερι. Εάν ναι, δεν έχει νόημα αυτή η ακρόαση. Σας ευχαριστώ. Οπότε ολοκληρώνουμε. Δεν είναι δύσκολο νομίζω να βγουν συμπεράσματα από την συζήτηση. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα το ξέπλυμα χρήματος μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κρίσιμο και εκρηκτικό θέμα. Ξεπερνάει τα οικονομικά εγκλήματα που συνήθως ε, συζητάμε και υπάρχει μια σοβαρή υποψία που συχνά βασίζεται και σε στοιχεία ότι τα χρήματα αυτά μπορεί να επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων σε κράτη-μέλη της Ένωσης, ε, να επηρεάζουν τις εκλογές, τα δημοψηφίσματα ή και το, κάποια επίπεδα δείξεις. Όταν μιλάμε για ξεπλήμα χρήματος, κάποια κράτη-μέλη είναι πιο ευάλωτα από άλλα και παίζουν μεγάλο ρόλο τα χρήματα εκεί. Πρέπει οπωσδήποτε να διευρύνουμε τα εργαλεία, τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας σε όλα τα επίπεδα για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την θεμελιώδη απειλή. Θα το κάνουμε στην έκθεσή μας, είμαι σίγουρος, από την σκοπιά του ξεπλήματος χρήματος και των σχετικών ζητημάτων και είμαι σίγουρος ότι η ακρόαση αυτή επίσης ε, βοήθησε στην ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα και την πολυπλοκότητά του. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους ομιλητές ε, για την συνεισφορά τους. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζεται η συνεδρία σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ξαναρχίσουμε τη συνεδρία της Επιτροπής ΤΑΞ 3 για να εξετάσουμε τις τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης. Θα ξεκινήσουμε με, τον, με τους συνεισηγητές. Θα δώσουμε πέντε λεφτά στον καθένα. Λούντεκ Μάγερ από το ΕΛΚ. Uh, uh, Μάλιστα. Ελπίζω να μην χρειαστώ και τα πέντε λεπτά. Μισό λεπτό. Καταρχάς, εκτιμώ τη δουλειά του συναδέλφου μου, του συνεισηγητή και των υπόλοιπων ε, σκιωδών και την υποστήριξη της γραμματείας γιατί είναι δύσκολο να ετοιμάσει κανείς μια τέτοια ε, έκθεση με 1.300 τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντική έκθεση αυτή, γιατί δεν αφορά μόνο αυτή την Επιτροπή, αλλά συνοψίζει όλη τη δουλειά που έχει κάνει το Κοινοβούλιο στον τομέα της, ε, του ξεπλήματος του χρήματος, δίκαιης φορολόγησης και των φορολογικών σκανδάλων. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μία από την ε, πιο σημαντικές οικονομικές εκθέσεις που έχει ετοιμάσει το Κοινοβούλιο. Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε μια έκθεση σοσιαλιστών και λαϊκού κόμματο. Θα συμφωνήσει και ο συνεισηγητή. Θέλω να ε, υπάρχει πραγματικά πλατή μέτωπο υπέρ τη έκθεση αυτή από όλε τι ομάδε, από όλου του βουλευτέ. Ε, φυσικά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι όλοι ενθουσιοδός υπέρ της ε, έκθεσης, αλλά με μεγάλη χαρά θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω όσο να το περισσότερες τροπολογίες και ελπίζω να το εκτιμήσετε αυτό. Και βασιζόμαστε σε αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Χρησιμοποίησαμε όσο μπορούμε τις, τα πορίσματα των ακροάσεων και ελπίζω τελικά να είναι μια φιλόδοξη έκθεση, μια καλή βάση για να συνεχίσουμε τη δουλειά αυτή για το θέμα αυτό στο μέλλον γιατί νομίζω ότι τα θέματα της δικής φορολόγησης, καταπολέμησης του οικονομικού και φορολογικού εγκλήματος και του ξεπλήματος του χρήματος είναι πάρα πολύ σημαντικά και τώρα και στο μέλλον. Είμαστε πολύ κοντά στην ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή. 27 Φεβρουαρίου θα λάβει χώρα. Στο μεταξύ όμως θα γίνουν πολλές συνεδριάσεις με τους συζητητές και χαιρετίζω την ε, εμπλοκή τους, στην συνεργασία τους, ε, στις ε, μέχρι τώρα δύο συνεδριάσεις. Έχουμε ε, συζητήσει τα 5 από τα 9 κεφάλαια. Στις επόμενες τρεις συνεδριάσεις θα έχουμε ε, διατρέξει όλη την έκθεση και θα ετοιμάσουμε συμβιβαστικές τροπολογίες που δεν θα αποκλείουν κανένα και καμία άποψη. Φυσικά το θέμα είναι οριζόντιο. Ε, κοινωνική διάσταση, ελάχιστη φορολόγηση, ε, κοινωνική διάσταση της ε, φορολόγησης, η φορολογική παράδειση που μπορούν να δημιουργήσουν ε, προβλήματα. Προσπαθούμε να φτιάξουμε όμως, ε, να χτίσουμε συνενέσεις, τουλάχιστον ε, σε κάποια σημεία του κειμένου και ελπίζω η καλή συνεργασία να συνεχίσει και τις επόμενες εβδομάδες και να ετοιμάσουμε μια έκθεση που θα μας κάνει περήφανος. Ευχαριστώ. Κλούντεκ. Ο κύριος Κοπ, από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Λούντεκ και τους συναδέλφους στην Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι δύσκολη δουλειά και θέλω να σας ευχαριστήσω τώρα ε, είπε ο Λούντεκ το πώς εργαστήκαμε. Γεγονός είναι ότι λάβαμε 1284 ε, τροπολογίες και πραγματικά νομίζω αυτό καταδεικνύει το πόσο σημαντικό θεωρούν τα μέλη της Επιτροπής ε, την δουλειά αυτής, της Επιτροπής αυτής της δικής μας αλλά και της Επιτροπής για τα έγγραφα του Παναμά και των άλλων δύο επιτροπών βεβαίως. Οπότε, να αναφέρω τις ε, αρχές μας εδώ πέρα. Ε, δεν ε, θα εγκρίνουμε και δεν θα προτείνουμε τροπολογίες που στόχο έχουν την διαγραφή την αποδυνάμωση του αρχικού κειμένου. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, προσπαθούμε να δεχτούμε σχετικά νούμερα και γεγονότα που ασίζονται σε αντικειμενικές πηγές ε, αρκεί να μην γίνονται επαναλήψεις βεβαίως. Ε, πρέπει να το πούμε αυτό. Ε, τι θέλουμε, να έχουμε καινούργια στοιχεία για να βελτιώσουμε την έκθεση. Τρίτον, θα τα ομαδοποιήσουμε τα των ομάδων και ένα θέμα. Οπότε αυτή την μεθοδολογία θα ακολουθήσουμε και από την πολιτική σκοπιά να πω ότι προχωράμε καλά, το είπε και ο Λοντέκ. Και βλέπω πως ε, υπάρχει επικοδομητικό πνεύμα στην αναζήτηση συμβιβασμών. Νομίζω πως η τελική έκθεση έχει αρκετή ουσία για να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο που δεν είναι αρκετά φιλόδοξο και συνεργάσιμο. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση λοιπόν στο Συμβούλιο στο τέλος της εντολής μας. Αλλά σας ε, διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενσωματώσουμε τις ε, τροπολογίες σας. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ, δεν θα εξαντλήσω τα πέντε λεπτά. Να πω ότι το πρόγραμμα είναι πιεστικό και πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί για να γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή όπως έχουμε προγραμματίσει. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ Γέπε. Προχωράμε. Λοιπόν, μόλις κότγεται για τους πράσινους. Έχω τελεθεί από τη χαρά μου, το βλέπετε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ τους συνεισηγητές ε, και το προσωπικό που εργάστηκε εδώ γιατί όπως είπε ο ΓΕΠΕ είναι πάρα πολλά τα θέματα αυτά και οι τροπολογίες. Έγραψα ένα tweet εγώ πριν την προηγούμενη συνεδρίαση γιατί ήταν χαοτική η κατάσταση και μιλάμε για μόνο δύο κόμματα με 12 χώρες ενώ την προηγούμενη φορά ήταν ε, πολύ χειρότερα τα πράγματα και ήμασταν πιο παραγωγικοί. Τέλος πάντων. Εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι ούτως ή άλλως με την έκθεση. Θεωρούμε ότι είναι ένα θετικό αποτέλεσμα της ε, δουλειάς της Επιτροπής μας. Της ε, πολλωστής ε, Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων. Και νομίζω ότι μετακινείται η πολιτική πλειοψηφία και θέλει πλέον ε, να αναλυφθεί κάποια σοβαρή θράση κατά της φοροαποφυγής, ε, φοροδιαφυγής και ξεπλήματος ε, χρήματος. Και για μένα είναι σαφές ότι και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να κάνουν τέτοιες έρευνες για να μην στέλνουν μετά κόσμο να τα μπλοκάρει αυτά στο Συμβούλιο. Γιατί όπως λέει ο Γέπε, εκεί κολλάμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους συνεισηγητές που περιέλαβαν πολλές τροπολογίες μας δεδομένου του ότι ήταν 1248 Χαίρομαι που πολλές δικές μας είναι στις ε, συμβαστικές ε, προτάσεις. Θεωρούμε ότι η έκκληση για διαφάνεια πρέπει να ενισχυθεί. Παραδείγματο χάρη πρέπει να δημοσιεύονται οι συνεδριάσεις της ομάδας επαφής ε, και οι χώρες εκείνες οι οποίες δεν συνεργάζονται. Ζητάμε επίση από τα κράτη-μέλη να υπολογίσουν ποιο είναι το κενό εκείνο της ε, φορολογίας για να έχουν κάποια κοινά κριτήρια αξιολόγησης του προβλήματος. Θεωρούμε ότι μπορεί να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία και να κλείσουν κάποια παραθυράκια στην, ε, που αναφέρουν στην έκθεση, αναφέρουμε εμείς οι πράσινοι στην έκθεσή μας. Ε, δεδομένου ότι πολλά από αυτά τα θέματα έχουν κολλήσει στο Συμβούλιο, θα ήθελα να επαναλάβω το ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική πλειοψηφία για τα φορολογικά και ελπίζουμε η Επιτροπή μας και το Κοινοβουλίο να τα ζητήσουν αυτά. Συμπερασματικά λοιπόν αναμένουμε την έγκριση πολλών τροπολογιών μας μεταξύ των οποίων αυτή που αναφέρει τις κοινωνικές συνέπειες της άδικης φορολογίας και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον κοινωνικό αντίκτυπο της φοροαποφυγής. Μία έκθεση της Oxfam την προηγούμενη εβδομάδα κατέστησε σαφή την σχέση του θέματος αυτού με την ανισότητα ε, και βεβαίως τα ζητήματα φορολογικής απάτης ε, και παράτυπων χρηματικών ροών. Και γνωρίζω βεβαίως πως εντάξει, όλοι εδώ πέρα έχουμε έναν κοινό στόχο να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών μας και να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να δουλέψουν λίγο και διερμηνείς, λες και δεν δουλεύανε τόση ώρα. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές. Πιστεύω ότι ακολουθεί τη γραμμή που έχουμε ορίσει και είναι και υποδειγματική η έκθεση ως προς τις επιλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον συγχρονισμό και την έκφραση σε όρους αυτού των θέσεών του που ταυτίζονται άλλωστε και με τις θέσεις και ανησυχίες των πολιτών, πολύ σημαντικό σε περίοδο προεκλογικής εκστρατείας. Είμαστε στην τρίτη ε, Επιτροπή για τη διερεύνηση των σκανδάλων ε, φόρου αποφυγής ε, και ιδιαίτερα νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο και συμβολικό χαρακτήρα η υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει το Κοινοβούλιο με την, ψηφοφορία, με την πρόταση για ψηφοφορία σε θέματα ε, φορολογικά ε, στο Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Πολύ σημαντικό για το μέλλον. Κάποιες παρατηρήσεις λοιπόν για να επαναλάβω ορισμένες προτεραιότητες. Η πρώτη και προς τους δύο συνεισηγητές ε, θέλω να απευθύνω το ερώτημα σε ποιο βαθμό και από ποιου όρους σκοπεύουν να λάβουν υπόψη τις εξελίξεις των εργασιών κυρίως του ΩΣΑ που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα όχι μόνο στο πλαίσιο του ΩΣΑ αλλά και αυτό που ονομάζεται «Inclusing Framework 177 χώρες μπορούν να παρέμβουν στην θεματολογία αυτή. Είχαμε πάντα αυτή την, αυτή την ευγενή άμυλα μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και όσα που είχε παρεμποδίσει σε κάποιο βαθμό τον ΩΣΑ, αλλά νομίζω ότι μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε κυρίως στην ψηφιακή φορολογία και την ε, θεώρηση του χώρου που θεωρείται σταθερή έδρα και βέβαια της ε, μεταφοράς κερδών στο ιστορικό ενός ομίλου. Αυτό το inclusion Framework έχει σημασία να το δούμε σήμερα, πρέπει να το λησμονήσουμε φυσικά. Αλλά βλέπουμε μια κινητικότητα η οποία όταν είχαν κατατεθεί οι τροπολογίες δεν είχε εκδηλωθεί και νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τρόπους και μέσα ώστε να προσαρμόσουμε το συντονισμό αυτής της έκθεσης και προς την αυτή εξέλιξη. Και δεύτερο σημείο αυτά που θα μπορούσαμε να, νομίσουμε, να ονομάσουμε πολυσυγκάπ. Δηλαδή, και το είπε και η Σκοτ Μόλι τώρα, ότι τα κράτη-μέλη αφήνουν κάποια χώρους φορολογικής ε, δραστηριοποίησης που μπορεί να μην χαρακτηρίζονται ως βελτιστοποίηση ή φοροαποφυγή, αλλά πάντως σημαίνουν ε, πολύ σημαντική συμβολή την δραστηριότητα του φορολογικού dumping. Υπάρχουν όμως νόμιμοι τρόποι ε, που έχουν στη θέση τους με βάση και την οδηγία του 2011, αν δεν απατώμε, τα κράτη-μέλη να ε, εντοπίσουν αλλά και να υπολογίσουν το κόστος αυτού του policy gap. Και ξέρω ότι μπορεί να ψάχνω ψήλου στα χειρά, αλλά η, 679 τροπολογία που αναφέρεται στα συμπεράσματα από το σκάνδαλο Κούμεξ ε, για τα όσα έγιναν. Ε. Εντάξει, εδώ στο Κοινοβούλιο όμως νομίζω μπορούμε να μην τα ανοιχτά. Δεν λέω ότι πρέπει να ε, δακτυλοδείχνουμε τον καθένα, να κάνουμε name and shame, αλλά να κάνουμε και λίγο name dropping, να πούμε και κανένα όνομα στα νύχτα. Έχει έρθει μπροστά μας μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες ε, μη συνεργαζόμενες ε, δικαιοδοσίες γιατί όταν αρχίζουμε τα μη μου απ' του άκεπο που μην πούμε τίποτα και μην το μάθουν τα παιδιά ε, δεν γίνεται τίποτα και μετά βγαίνουμε προς τα έξω για να ζητήσουμε κάτι, να προβάλλουμε κάποιες θέσεις και ο ψηφοφόρος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ακόμα και ο δημοσιογράφος δεν καταλαβαίνει μερικές φορές. Έτσι λοιπόν, για να μου δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο κύριε Πρόεδρε, ε, αυτή η συζήτηση που ξέρουμε ότι θα στρώσει και τις εργασίες μας εν ώψη του προσεχούς ε, κοινοβουλίου όταν θα υπάρχει υποεπιτροπή μόνιμη ή όχι πρέπει να είμαστε απόλυτα ε, αποφασισμένοι αντί της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής και αυτό το λέω όχι μόνο γιατί είμαι μέλος των δύο αυτών επιτροπών αλλά και γιατί πιστεύω και η τελευταία μου αυτή παρατήρηση ε, επιρρονεί τα όσα έχω να πω ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα θέματα αυτά δεν μπορούμε να αποκόψουμε τα θέματα αυτά από την οικονομική και νομισματική ιδάλω. αποκόπτουμε τα φορολογικά θέματα από τη λειτουργία των αγορών. Άρα είτε πρόκειται για κίνητρα, είτε πρόκειται για έλεγχο και κυρώσεις, χρειάζεται αυτός ο σύνδεσμος και φτάνω στη τελευταία μου παρατήρηση. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει καλύψει η έκθεση και άρα δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το ε, συμπληρώσουμε όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι αρχές δηλαδή οι οποίες αυτή τη στιγμή εξετάζουν, μελετούν ε, το σκάνδαλο Κούμεξ και πάνω απ' όλα τη λειτουργία και την εποπτεία των αγορών, αυτές οι αρχές δεν έχουν τώρα το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν φορολογικά δεδομένα που συλλέγουν οι φορολογικές αρχές. Τεράστιο κενό προφανέστατη έλλειψη στα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους αυτές οι αρχές εποπτείας για εντοπισμό των κενών στο διατακτικό και άρα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει η έκθεσή μας γιατί είναι και πολύ επίκαιρο. Πρόεδρε, υποπτεύομαι ότι μακρηγόρησα κάπως αλλά ήθελα οπωσδήποτε να επισημάνω τα σημεία αυτά για τους δύο εισηγητές στους οποίους εύχομαι και πολύ καλή τύχη για την ολοκλήρωση της έκθεσης. Ευχαριστώ. Τάνκ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους ε, εισηγητές για τη δουλειά τους. Ε, πολλά υποσχόμενη έκθεση. Υπάρχουν βέβαια και πολλές τροπολογίες. Τώρα το συνειδητοποίησα. Καλή τύχη και καλή δύναμη. Καλή εντύπωση έχω. Όπως και η ε, θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι μπορούμε να στείλουμε δύο μηνύματα. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε μια ενιαία θέση, αλλά και εν ώψη προεκλογικής εκστρατείας δεν θα πρέπει να αποφύγουμε να παρουσιάσουμε τις διαφορετικές απόψεις, γιατί πολιτικό όργανο είμαστε, διαφορετικές απόψεις κυκλοφορούν εδώ. Δεν θα πρέπει να έχουμε πρόβλημα με αυτό. Κοιτώντας τελευταία περίοδο, βλέπουμε μια ελληματική Ευρώπη. Μπορούμε να αφισβητήσουμε την ικανότητα της Ευρώπης να κάνει διαφορετικές αλλαγές στη φορολογία. Ειδικά μια τέτοια μέρα που ο ΣΑ κάνει πιο φιλόδοξες προτάσεις ε, για τον DST, από το, το DST που ήταν πάντα προσωρινό και έχει αποκλιμακωθεί, αποδυναμωθεί κτλ. Εμείς τι δείχνουμε, ότι είμαστε διαιρεμένοι. Το θέμα είναι λοιπόν τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε ως Ευρώπη. Εάν θέλουμε να παίξουμε κάποιο ρόλο θα πρέπει να ενωθούμε και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το γεγονός ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί, ευρωπαίοι εταίροι που ε, λειτουργούν εις βάρος άλλων ευρωπαίων εταίρων. Θα πρέπει να τα καταγγέλουμε αυτά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, θα πρέπει να λέμε ποιες χώρες μπλοκάρουν τη διαδικασία. Δεν θέλω τώρα να στυλιτεύσω συγκεκριμένους, αλλά νομίζω ότι αυτό μπλοκάρει την ευρωπαϊκή προσέγγιση τώρα, ειδικά που έχουμε και την διεθνή συζήτηση, η οποία είναι ανοιχτή, είναι σημαντικό να παίξει το ρόλο της η Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και τη δουλειά που έχει κάνει ο και να δούμε αν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή έχουμε θέσεις, ειδικά για το CCTB, ε, που αλλάζει πολύ τα δεδομένα του παιχνιδιού και τη συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά έχουμε και, σημαντική, και το νομοθέτημα για τη σημαντική ψηφιακή παρουσία. Είναι νομοθέτημα το οποίο έχει στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε αυτά να τα προτάξουμε για να δείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε ενιαίο μέτωπο στη συζήτηση του ΩΣΑ για να φωτίσουμε και το δρόμο προ τα εμπρό. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι όλοι οι βουλευτέ που είναι παρόντε μίλησαν. Ξαναδίνω το λόγο στου εισηγητέ. Ο Λούντικ πρώτο. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Για τον ΩΣΑ Σήμερα εκδόθηκαν κάποια κείμενα. Θα το εξετάσουμε το κείμενο αυτό πολύ προσεκτικά, γιατί όσα είναι μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές για μας. Συμφωνώ με αυτό που ακούσαμε. Φυσικά θα υπάρξουν πολιτικές διαφορές, αλλά σε τομείς όπου μπορούμε να συμφωνήσουμε, ε, θα προσπαθήσω και το προτιμώ να βρω συμβιβασμούς. Φυσικά θα υπάρξουν λοιπόν διαφορές, αλλά εκεί που μπορούμε να βρούμε ένα καλό κείμενο αποδεκτό είναι προτιμότερο βεβαίως. Αυτά ευχαριστώ. Γεπέντ, ευχαριστώ. Ναι, προς την μόλη. Κάποιες ε, τροπολογίες ε, αναφέρουν συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς ε, που πρέπει να μπουν στην έκδοση και αποτελούν την βάση της ε, έκθεσής μας. Ε, λοιπόν, για τη σημερινή πρόταση του ΩΣΑ, χωρίς την ευρωπαϊκή συζήτηση δεν θα είχε κινηθεί ο ΩΣΑ. Οπότε πρέπει να αναγνωρίσουμε και τον ρόλο που παίξαμε κι εμείς. όσον αφορά ακριβώς ε, την δίκαιη εταιρική φορολογία. Ε, και τώρα βεβαίως αναζητάμε ένα BEPS 2 ε, και μετά για τις χώρες της Ένωσης. Είναι σαφές ότι έχουμε πολιτικές διαφορές, αλλά από τη δικιά μου σκοπιά νομίζω είναι σημαντικό ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένωση με βέτο ή δικαίωμα του κράτους μέλους να υπονομεύει την δουλειά που γίνεται κατά των ε, βλαβερών διασυνοριακών ε, φορολογικών καθεστώτων. Είναι σαφές. Και αυτό πρέπει να το πάμε και στην ε, Ολομέλεια. Να πούμε δηλαδή τουλάχιστον ότι η αρχή της ομοφωνίας ε, προστατεύει τους ε, ευρωπαϊκούς φορολογικούς ε, παραδείσους. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε σε τέτοια ζητήματα ειδική να έχουμε βέτο, πρέπει να περάσουμε σε μια ειδική πλειοψηφία, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και βεβαίω ε, και από την σκοπιά του ανταγωνισμού, ο οποίο πρέπει να είναι πιο δίκαιο. Αυτά λοιπόν, Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμένουμε κι εμεί προσεχώ να σα πούμε το τι έγινε με τι ε, συμβιβαστικέ ε, τροπολογίε. Σα ευχαριστώ. Η ψηφοφορία είναι στι 27 Φεβρουαρίου το πρωί και θα ψηφίσουμε πιθανότατα στη δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όσους έμειναν μέχρι τώρα. Η επόμενη συνεδρίαση στις 4 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και τους ερμηνείς. Αυτά για σήμερα.